Κυρίε και κύριοι, ε, ξεκινάει η συνεδρίμασή μας ε, για σήμερα το απόγευμα. Οι ε, ψηφοφορία σήμερα το πρωί ήταν τόσο κουραστικέ ώστε ορισμένοι έχουν παρατείνει το μεσημεριανό διάλειμμα για να συνέλθουν αλλά έχουμε εδώ την, την Πία Λοκατέλη με μια ομάδα μαθητών από την Ιταλία τους οποίους καλωσορίζω στην Επιτροπή μας και για το ενδιαφέρον για την εργασία μας και βρισκόμαστε στο σημείο 12 δραστηριότητες της ΣΤΟΑ σχετικά με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. και εδώ συγκεκριμένα ε, στην ΣΤΟΑ που σημαίνει Science and Technology Assessment ε, Έχουμε ε, δύο εκπροσώπους, τον κύριο Πρόντι από τους σοσιαλιστές και έναν εκπρόσωπο από, τους, ε, από το ΕΛ ε, οι οποίοι θα μας πούν τι μπορούμε να κάνουμε με τα διάφορα θέματα τα οποία παρακολουθούμε. Και θα δώσω στον κύριο Ταταρέλα τον λόγο για να κάνει την πρώτη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ιδιαίτερα για αυτή την πρώτη συνάντηση, αυτή την πρώτη δυνατότητα που έχουμε εμείς ως μέλη της ΤΟΑ να, σας, ε, ε, να αναφερθούμε στις δραστηριότητες μας και να σας καταδείξουμε τι ακριβώς έχουμε επιτύχει. Γιατί από όσο γνωρίζω, σε καμία άλλη παρόμοια επιτροπή δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ ΣΤΟΑ και Κομισιόν θα πρέπει να ενδυναμωθεί έτσι ώστε η δραστηριότητα της ε, ΣΤΟΑ να αποτελέσει αντικείμενο συσχετισμού εργασιών με τις επιτροπές. Φτάνουν στη ΣΤΟΑ πολλά προσχέδια προγραμμάτων και δεν θα ήταν σωστό η ΣΤΟΑ να αποφασίσει χωρίς να έχει επαφή με τις επιτροπές αναφορά. Σας ευχαριστώ λοιπόν, διότι η η πρώτη επιτροπή που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Τα προγράμματα δεν επιλέγονται τυχαία. Γίνεται μια εσωτερική αξιολόγηση και νομίζω ότι εδώ για πρώτη φορά σε μια πρόσφατη συνεδρίαση της 20ης Μαΐου τα προγράμματα ψηφίστηκαν. Άρα ως Επιτροπή ΣΤΟΑ επιλέξαμε τα σχέδια που ε, θα μας απασχολήσουν. Θα σας ε, δώσω έναν απογραφικό κατάλογο μαζί με τον συνάδελφο Βιτόριο Πρόντι. Και αρχίζω με ένα καλό νέο. Το πρόγραμμα που υπερψηφίστηκε κατά πολύ είναι το πρόγραμμα ΕΝΒΗ για την αηφόρο ανάπτυξη των υδάτων που έτυχε ευρύτατη συνένεσης. Ένα δεύτερο σημαντικό πρόγραμμα είναι εκείνο που υπέβαλε ο πρόεδρος ε, του ΣΤΟΑ, ο κύριος Ρούμπιχ, και αφορά τις απειλές κλιματικών αλλαγών και τις επιπτώσεις στη γεωργία που όπως γνωρίζουμε είναι υπεύθυνη για το 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ένα τρίτο project έχει ως αντικείμενο τη σημασία της αστρονομίας και τη νέα χαρτογράφηση του πλανήτη. Πρόκειται για ε, ένα workshop το οποίο ε, συμφωνήθηκε και από τον κύριο Μαντουρέλ. Υποστηρίζουμε την ε, σημασία της αστρονομίας, την αστρονομία κάθε αυτή, καθώς και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ως προς τα αποτελέσματα των εκπομπών στο διάστημα. Θα πρέπει να δούμε τα, τις νέες πηγές ενέργειας, τις, ε, τη νέα αντιμετώπιση και θεραπείες και τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς και τις μεταφορές στο γεωργικό τομέα. Ένα άλλο πρόγραμμα αφορά όχι μόνο τη δική μας Επιτροπή, αλλά και την Επιτροπή Μεταφορών και την Ήτρε αφορά την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων στο ενεργειακό σύστημα. Το θέμα των ηλεκτρικών οχημάτων, των κινητήρων και την αυτοκινητοβιομηχανία δίνοντας σημασία στη διατηρήση θέσεων απασχόλησης. Επίσης συμμετέχω και σε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι ύψης της σημασίας για τις εργασίες μας. Θέλαμε να συνοδεύσουμε τις εργασίες του Κοινοβουλίου με το κόσμο και τις επιστήμης, έτσι ώστε να υπάρχει αυτός ο άλληλος συσχετισμός μεταξύ ε, επιστήμης και κοινοβουλευτικών εργασιών. Ένα τελευταίο θέμα αφορά το Smart Grid για την ενέργεια, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να δούμε τις ανανεώσιμες πηγές και να βοηθήσουμε για τις ε, παράπλευρες υπηρεσίες, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να ελέγχουμε αυτά τα ευφύ συστήματα. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρόντι. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας ε, είπατε. Και ε, τώρα ο κύριος ε, Πρόντι έχει το λόγο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Συμφωνώ με το συνάδελφο Ταταρέλα, διότι αναφερόμαστε στις ε, εργασίες της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος σε σχέση με τις εργασίες της ΣΤΟΑ. Σημαίνει στήλη, λέει ο κύριος πρώτη στα ελληνικά, λάθος. διότι δεν μιλάμε για παράπλευρα ζητήματα. Τι σημαίνει, σημαίνει πυλώνας, κολώνα, τι. Uh, uh, Είναι κάτι που υπάρχει στα ορυχεία, μια στοά δηλαδή που υπάρχει στα ορυχεία. <laughs> για τη διέλευση σε αυτά. Mind. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Πρώτη. Ε, είναι οι γνώσεις μου από το Λύκειο, όπως καταλαβαίνετε. Κατανοείτε τι αξία έχουν. Εν πάση περιπτώσει, θυμόμουν ότι είναι κάποιο στοιχείο, κάτι, ένα κατασκευαστικό στοιχείο, ένα στοιχείο κατασκευών. Υπ' αυτή την έννοια ε, χαίρομαι για τη διευκρίνηση. Το θέμα, μάλλον η ενιολογική βάση βασίζεται στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία κοινωνία τάχιστων εξελίξεων και έχουμε νέες επιλογές οι οποίες απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες, αλλά και από την προώθηση του, του, της ε, επιστήμης και την εξέλιξη της επιστήμης. Για παράδειγμα, όλοι αντιμετωπίσαμε την αρχή της ε, προστασίας την αρχή της προστασίας και την, και ανάγκη να κατανοήσουμε πώς η αρχή της έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πώς θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν τελικές οριστικές γνώσεις τις οποίες να συμμερίζονται όλοι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην αναλάβουμε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να έχουν ε, απρόβλεπτες συνέπειες. Επειδή ακριβώς αναγνωρίζουμε ότι είναι περιορισμένες οι γνώσεις μας, θα πρέπει αυτή τη φάση να την υπερβούμε το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να έχουμε επαρκείς γνώσεις για να περάσουμε από την αρχή της πρόληψης των προληπτικών μέτρων σε μία αποτίμηση κινδύνου, ποσοτικού κινδύνου. Διότι πολύ συχνά Χρησιμοποίησαμε αυτή την αρχή της πρόληψης για την ε, ε, ανάληψη δράσης. Η ΣΤΟΑ λοιπόν προσπαθεί να υποστηρίξει και τη δράση του Κοινοβουλίου προς τη μεθοδολογία για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα τα οποία μπορεί να είναι τεχνολογικά ή πολιτικά, τεχνολογικής ή πολιτικής φύσης. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε στη διάθεση του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα, να αντιμετωπίσουν ορισμένα προβλήματα. Ο κύριος Ταταρέλα μίλησε για θέματα τα οποία έχουμε αναλάβει ως προς το πρόγραμμα εργασίας της ΣΤΟΑ και βεβαίως όλα αυτά αφορούν μία γενικότερη συλλογιστική που μας διέπει στον τομέα της ενέργειας, της γεωργίας και θα ήθελα να δούμε τα όρια μας ως προς τους φυσικούς πόρους. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να οριοθετήσουμε αυτή την κατάσταση και τι επακριβώς σημαίνει. Ζούμε σε έναν πολιτισμό ο οποίος δεν γνωρίζει αυτά τα όρια, γιατί για πολλά χρόνια το ανθρώπινο είδος γνώριζε πρωτόγονες τεχνολογίες ή τεχνικές. Τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση όπου βλέπουμε πώς έχει αυτός ο διτός περιορισμός με βάση την πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε και να προσπαθήσουμε να συνοδεύσουμε αυτή την ε, τεχνολογική εξέλιξη, τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσα στα πλαίσια μιας εύλογης ασφάλειας ως προς τη, τους διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε κατάσταση έλλειψης πόρων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα κινητό απαρτίζεται από 30 ε, στοιχεία. Ε, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία είναι σπάνια. Έχουν ένα δείκτη σπανιότητας ή σπάνιδος. Ε, άρα η αρχή του, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν αφορά θέμα μόνο αποβλήτων αλλά και θέμα πόρων. θα πρέπει να ορίσουμε αυτούς τους όρους που θα πρέπει να μας διέπουν σε όλες τις αποφάσεις. Η ΣΤΟΑ λοιπόν προσπαθεί να δώσει απαντήσεις μέσα στα πλαίσια των νανοτεχνολογιών θέλουμε να δώσουμε εναλλακτικέ σε υλικά τα οποία είναι αναντικατάστατα ή σπάνια υλικά σε σχέση με τα κοινότερα, τα οποία χρησιμοποιούμε με σύνεση. Από τεχνολογικής πλευράς, όπως τους νανοαγωγούς, από, ε, ε, στοιχεία από άνθρακα και ούτω καθεξής. Υπάρχει μεγάλος υψηλός βαθμός περιπλοκότητας δηλαδή και υπάρχουν και οι τοξικολογικές μελέτες στα πλαίσια της νανοτεχνολογίας γιατί για τα ε, μόρια αυτά, αυτά τα νανομόρια θα μπορούσαν, μπορούν να παρουσιάζουν διαφορετική τοξικολογία από αυτή που γνωρίζουμε. Αυτά τα μικροσωματίδια τα νανοσωματίδια δηλαδή ίσως μπορούν να μπουν απευθεία στο κύτταρο χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς πώς. μέσα στα πλαίσια και της ε, βιομηχανικής. Υπάρχει βέβαια και θέμα δεοντολογίας που σχετίζεται άμεσα με αυτά τα δεδομένα, με τη χρήση δηλαδή της βιοτεχνολογίας ή της μηχανικής. Άρα αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική διότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος μπορεί να κατανοήσει πού μπορεί να στηρίξει την ομάδα ΣΤΟΑ ως προς τη δυνατότητα απορρόφησης και απόφασης, λήψης αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόντι. Χαιρετίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση διότι αναφυσβήτητα η Επιτροπή στο είναι σημαντική για την Επιτροπή Περιβάλλοντος όπως και για άλλες που αντιμετωπίζουν περίπλοκα θέματα όπου οι μελέτες της Επιτροπής ΣΤΟΑ μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε, στη σωστή ε, αξιολόγηση. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε αν χρησιμοποιούμε παρκώς την Επιτροπή ΣΤΟΑ ή ε, αναπαρκώς. Και αυτό εγκαίρως προτού προχωρήσουμε προς τη λήψη αποφάσεων και στις ψηφοφορίες. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίζουμε ε, διότι αναφερόμαστε σε θέματα σχετικά με τη χημεία, με τη βιολογία που δεν τα έχουν σπουδάσει όλοι και πολλές φορές είναι περίπλοκο να γνωρίζει ακριβώς τι επιπτώσεις υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχει η Επιτροπή ΣΤΟΑ. Όλα τα κοινοβούλια έχουν μια Επιτροπή σαν τη ΣΤΟΑ. Το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει την πιο σημαντική ε, επιστημονική υπηρεσία και γι' αυτό εμείς είμαστε ευγνώμονες στην Επιτροπή ΣΤΟΑ η οποία εκτός από τις ε, ε, και ιδίως τους συναδέλφους οι οποίοι εκτός των όλων καθηκόντων τους ασχολούνται και με αυτή την Επιτροπή. Ε, δεν ξέρω εάν κάποιος ε, έχει κάποια ερώτηση διότι ενδεχομένως ε, ε, κάποιος ε, θέλει ε, να σχολιάσει αν εργάζεται υποπίεση ή ελεύθερα. Επίσης θα ήθελα να ξέρω εάν οι μελέτες γίνονται από δικούς μας ανθρώπους ή υπάρχει υπεργολαβία και αναθέτουμε έξω τις μελέτες αυτές. Επίσης χαιρετίζω ιδιαίτερα στο ότι κάνουμε αξιολόγηση κινδύνων risk assessment διότι είναι μία ανησυχία μας και εγώ θα έλεγα ότι η Επιτροπή μας θα έπρεπε να συζητήσει γενικώς ε, ε, ε, τι, τι κίνδυνοι ε, ε, πώς γίνονται αντιληπτοί οι κίνδυνοι διότι οι πολιτικοί έχουν διαφορετική αντίληψη του κινδύνου από ότι οι τεχνοκράτες και ο κύριος Πρόντι είπε ότι πολλές φορές εμείς αποφασίζουμε να μην εγκρίνουμε κάτι το, για το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι καλό ή κακό ενώ επιστήμονες θα μπορούσαν να πούνε είναι παρκώς καλό, άρα μπορεί να το πράξει η βιομηχανία, αλλά κατά τη θητεία μας αυτή καλό θα ήταν να γίνει ένα εργαστήριο όπου να συζητήσουμε το risk assessment, να δούμε ακόμη τα περιθώρια που έχουμε για τη λήψη αποφάσεων και μετά να λάβουμε μία απόφαση. Ο κύριος Ταταρέλα έφυξε και ένα-δύο θέματα, δηλαδή τις επιχειρήσεις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών στη γεωργία και τις επιπτώσεις της γεωργίας στις κλιματολογικές αλλαγές. Όπως βλέπετε υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος και είναι βασικό να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Είναι μετά όσον αφορά ε, ε, το ε, νερό. Η Επιτροπή θα εκπονήσει μία στρατηγική για το νερό η οποία χρειάζεται από την Επιτροπή. Έχουμε επίσης ε, πολύ έμπειρους ανθρώπους εδώ, η κυρία Μεγέ, η οποία θα μπορούσε να τοποθετηθεί, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν επιθυμεί μπορεί να σχολιάσει την εργασία της Επιτροπής ΣΤΟΑ ή κάποιος άλλος. Αλλά αν δεν υπάρχει κανείς ενδιαφερόμενος, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε. Θέλω να ρωτήσω του συναδέλφους μήπως κάποιος, ε, θέλει, ε, θέλει να μιλήσει. Η Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε αλλά χάνω τη φωνή μου αργά και σταθερά. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σαν ευρωβουλευτές, να καθορίζουμε δημόσιες πολιτικές και να αξιολογούμε τα αποτελέσματα των πολιτικών τις οποίες έχουμε ε, καταρτήσει εάν δεν ε, έχουμε μία κοινή βάση αξιολογήσεως. Άρα, ό,τι μπορεί να γίνει για να ε, προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τις ε, συνθήκες υπό τις οποίες ε, βρίσκουμε αυτά τα στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο μας επικοινωνούνται είναι πολύ βασικό. Θα επανέλθω επίσης σε αυτό που είπε ο κύριος Πρόντι όσον αφορά την αρχή της ε, προφυλάξεως, της προλήψεως διότι βλέπω ότι αυτή τη στιγμή αμφισβητείται και αμφισβητείται καταρχήν γιατί γιατί ε, θα, ορισμένοι θεωρούν ότι χρειάζεται μία αρχή διαχείρισης του κινδύνου και όχι αξιολόγησης του κινδύνου ενώ εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται και τα δύο και παραπέμπω εις ε, την έκθεση πριν 10 χρόνια του οργανισμού ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όπου όλα αυτά εξηγόντουσαν πάρα πολύ καλά. Πέραν αυτού όμως η αμφισβήτηση της αρχής των προφυλάξεων προέρχεται διότι είναι πολύ αποστασιμοποιημένη η αρχή αυτή από την έρευνα. Η προφύλαξη είναι απλώς πλέον ένα θέμα δράσης ή αδρανίας ενώ θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό. Είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει όταν όπως είπε ο κύριος Πρόντι αντιμετωπίζουμε μη αποδεδειγμένους κινδύνους ε, πρέπει κανείς ε, να ε, ξεχωρίσει την προφύλαξη από την πρόληψη διότι όταν υπάρχει ένας μη αποδεδειγμένος ο κίνδυνος θα πρέπει να εμβαθύνουμε την έρευνα να θέσουμε τις σωστές ερωτήσεις για να υπάρξει μία επιτάχυση της έρευνας προτού φτάσουμε στο στοιχείο της πρόληψης δηλαδή υπάρχουν επιστημονικοί οργανισμοί οποίοι μπορούν να κινητοποιηθούν και να απαντήσουν στα ερωτήματα που μπορούμε να τους θέσουμε. Η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι ε, στο εάν ήδη μπορεί να ε, τεθούν οι ερωτήσεις διότι πρόκειται για θέματα τα οποία μπορεί να καταλήξουν σε αρνητικές απαντήσεις και σκέφτομαι παραδείγματος χάρη στις ε, γενετικές επιπτώσεις των τροποποιημένων οργανισμών και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ βασική. Ευχαριστώ κυρία Λεπάζ, σας εύχομαι ε, ανάρρωση διότι αντιλαμβάνουμε ότι στο Παρίσι δεν σας έκανε καλό η παραμονή στο συνέδριο. Νομίζω πως ε, άφησαν οι συνάδελφοι, δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος ε, τον λόγο, οπότε αν μπορείτε να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακούστηκαν ε, από το βήμα, ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, ο κύριος Πρόντι πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τις έρευνες γενικότερα, Οι έρευνες ανατίθενται προς τα έξω. Γίνεται εξωτερική ανάθεση, outsourcing. Διότι πολλές φορές εμείς δεν διαθέτουμε τις κατάλληλες ε, γνώσεις. Γι' αυτό θα πρέπει ακριβώς να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή επιστημονική ε, αρρωγή και υποβοήθηση. Το προσωπικό που αναλαμβάνει αυτή την διεργασία και βοηθά την Κομισιόν μπορεί ε, πάντα να είναι στη διάθεση όλων. Μας ενδιαφέρουν και οι δημοσιεύσεις της ΤΟΑ. και υποδείξεις Αυτό που έχει σημασία είναι να ληφθεί μία απόφαση η οποία να μην επιβληθεί τα έγγραφα αυτά παρουσιάζουν μία πληρότητα συνήθως. Με βάση τις ε, προσδοκίες μας βέβαια. Για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά. Υπ' αυτή την έννοια Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένα σωστό επίπεδο παροχής ε, συμβουλών, consulting, για να είμαστε σίγουροι για την εγκυρότητα της απόφασής μας. Αυτό απασχολεί όλους τους συναδέλφους της ε, ΣΤΟΑ. Δηλαδή να περιλάβουμε στο κείμενό μας, στα κείμενά μας, τις ε, καλύτερες ε, δυνατές γνώσεις, καθώς και τα ποσοτικά στοιχεία, αν λάβουμε υπόψη την αποτίμηση κινδύνων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να προβούμε σε αντιπαραβολές εκεί που χρειάζεται. και να έχουμε και μία δυνατότητα επιλογής. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος άλλος θα ήθελε να μας πει περισσότερα από το προσωπικό ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω σε όσα προελέχθησαν ότι ο προϋπολογισμός για φέτος είναι 150.000 ευρώ, λέει ο μιλητής, δηλαδή λίγο υψηλότερος. Θα πρέπει να πω με αυτοπεποίθηση ότι είναι ανεπαρκέστατος ο προϋπολογισμός σε σχέση με τους στόχους ε, του ΣΤΟΑ. διότι παντού και πάντα λέμε ότι η πόροι προς την έρευνα είναι ανεπαρκέστατοι. Εάν λοιπόν θέλουμε εμείς να μας βοηθήσει το ΣΤΟΑ, θα πρέπει εμείς πρώτοι να εφαρμόσουμε αυτό που επιβάλλουμε και σε άλλους. Δηλαδή, να αυξηθούν τα κονδύλια για τη ΣΤΟΑ. Ως προς τις εργασίες της ΣΤΟΑ, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι βασιζόμαστε σε εξωτερικά κέντρα ερευνών και πανεπιστήμια. Αλλά υπάρχει πάντα ένας υπάλληλος της Επιτροπής και ένας βουλευτής που στο μέτρο του δυνατού και των γνώσεών του προσπαθεί να βοηθήσει. Δηλαδή να προβεί σε ένα πολιτικό έλεγχο των εργασιών Και τέλος, αυτά τα στοιχεία δημοσιεύονται στο site μας, στην ιστοσελίδα μας. Το site της ΣΤΟΑ ε, θα πρέπει να είναι επικοδομητικό. Όχι μόνο από το Κοινοβούλιο, αλλά και από μια ευρύτερη κοινότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο δελεαστική η ιστοσελίδα μας και πιο εύκολα αναγνώσιμη. Έτσι ώστε ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα. Ευχαριστώ πολύ τους εκπροσώπους μας στην ΣΤΟΑ. Βεβαίως ε, η πύλη στο ίντερνετ είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα και στο μέλλον. Ελπίζω λοιπόν να είναι προσβάσιμη για το κοινό και όχι μόνο για κάποιους επιστήμονες, αλλά εάν όχι είναι και αυτό κάτι που πρέπει να αναφέρουμε στη πρακτικά αυτής της ε, συνεδρίασης. Επίσης θα ήθελα με την βοήθειά σας να κάνουμε ένα εργοστάσιο για την αξιολόγηση κινδύνου, για την ε, φιλοσοφία κινδύνου της Επιτροπής μας, αυτό το οποίο είπε η κυρία Λεπάζο, ο κύριος Πρόντι. Έτσι, δύο ρίτσες να μιλήσουμε σοβαρά για το τι είναι, ποια είναι η φιλοσοφία κινδύνου και ποια είναι η έννοια του κινδύνου με την οποία εργαζόμαστε. Οπότε σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας είπατε. Εύχομαι καλή επιτυχία. Υπερνάμε σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ε, στρατηγικής της βιοπικιλότητας και προοπτικές για τη νέα προοπτική της ε, βιοπικιλότητα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ντελάν και η οποία έχει εργαστεί μακρόν του θέματος και της δυνατολόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ειλικρινά πως ε, εργαστικά επ' αυτής της έκθεσης σκεπτόμενοι τον πατέρα μου, όχι γιατί είναι βιολόγος, είναι δάσκαλος γερμανικών και η αγαπημένη του παροιμία ήταν ε, ο καλός ο καπετάνιος στη φορτούνα φαίνεται, στα δύσκολα φαίνεται και βεβαίως με τους περιορισμούς που έχω εδώ πέρα βεβαίως θα έλεγε για το μην αναβάλεις για αύριο ότι μπορείς να κάνεις σήμερα και αυτό και αυτό Λοιπόν, ε, οπότε πράγματι εδώ πέρα πρέπει να είμαστε καπετάνιοι στα δύσκολα και στους πολλούς περιορισμούς που έχουμε γιατί η έκθεση είχε διπλάσιο ε, μήκος ε, αρχικά και βεβαίως μου είπε η γραμματεία πως πρέπει να περιορίσω τις σελίδες, τις παραγράφους ακόμα και τις λέξεις τον αριθμό των λέξεων. Οπότε περιοριστήκαμε στα βασικά και αυτά είναι τα οποία βλέπετε. Ο πυρήνας, δηλαδή η βάση, βρίσκεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια διεθνής ε, παράγραφος, αλλά βεβαίως αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα τελείω ξεχωριστό ψήφισμα διεθνές για την ε, Ναγκόγια, οπότε προσπάθησα να αναφερθώ κατά βάση στα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε όταν μιλάμε για τα Βασικά έχουμε την απογοήτευση για τη μη τήρηση του στόχου 2010, την ανησυχία που έχουμε για την μεγάλη ταχύτητα απώλειας της βιοπικιλότητας και το τι κάνουμε τώρα από εδώ και μπρο. Και πρέπει να σκεφτούν οι συνάδελφοι πώ πρέπει να σταματήσουμε την απώλεια τη βιοπικιλότητας και αυτό είναι ο ελάχιστος στόχο. και πρέπει να οδηγηθούμε προ μια αποκατάσταση. Να δούμε δηλαδή τι θα ε, γίνει γιατί αυτό ε, συχνά είναι απαραίτητο για να σταματήσει η απώλεια της ε, βιοποικιλότητας. Πολλές χώρες το κάνουν, οπότε πρέπει να παραμείνει στόχος στη μελλοντική στρατηγική η αποκατάσταση. Νομίζω αυτό πρέπει να το αναφέρει και η αξιολόγηση αντικτύπου. Και ένα τρίτο σημείο βεβαίως ε, είναι διεθνή ο χαρακτήρας του θέματος, οπότε αυτό σημαίνει πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει οι απόπειρε όλα αυτά τα οποία κάνει, να τα φέρει και σε ένα διεθνές επίπεδο, να τεθούν διεθνώς και να το προωθήσει αυτό περισσότερο. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να δούμε την επιλογή 4 στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως, όταν περιοριζόμαστε στα βασικά, αυτό σημαίνει πως δεν θα αναφερθούμε σε επιλογές οι οποίες γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών και αφορούν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτό βεβαίω αφορά την Natura 2000, καθώς στη δικιά μου τη χώρα υπάρχει μεγάλη αναταραχή για αυτή την πολιτική, το πώς λειτουργεί, τι αντίκτυπο έχει. 8-9 στις 10 φορές μιλάμε βεβαίως για αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί τελικά σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το κάνω όμως αυτό για 27 χώρες. Προσπάθησα να αναφέρω κάποιες μεγάλες διαφορές όπως τις βλέπω εγώ τουλάχιστον. Νομίζω και αυτό είναι καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη το ότι Κάποιες ε, χώρες ε, εξαιρούν ε, ολόκληρους τομείς από τον αρνητικό αντίκτυπο ενώ άλλες, που έχουν στη φύση ενώ άλλες δεν το κάνουν καθόλου, κάτι το οποίο προκαλεί εντύπωση. Επίσης ε, είναι ένα άλλο θέμα νομικό, δηλαδή όταν μιλάμε για το Natura 2000 είναι πάρα πολλές οι εθνικές αλλά και πάρα πολλές οι ευρωπαϊκές διατάξεις και αν δούμε ποιες είναι οι διατάξεις και οι αποφάσεις βλέπουμε πως η νομική εφαρμογή του τι σημαίνει το Natura 2000 είναι και αυτή συχνά διαφορετική. Δηλαδή εγώ είδα αποφάσεις ε, δικαστηρίων που έλεγαν πως δεν υπάρχει καμία απόφαση ε, αρνητικών αποφάσεων και είδα και δικαστές που λένε όχι εγώ θέλω αποδείξεις μη αρνητικών αποτελεσμάτων. Και βεβαίως ε, μιλάμε για τελείως διαφορετικό βάρος της αποδείξεως, οπότε Πρέπει να δούμε τι γίνεται βέβαια και με την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και με το, την εφαρμογή που έχει αυτή η νομοθεσία στο εθνικό επίπεδο. Και εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε μια όθηση. Τώρα ως ε, Ευρωπαία επίσης βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι σε κάποιες διασυνοριακές ε, περιοχές ε, περιοχές προστασίας οι οποίες διασχίζονται από ένα σύνορο δεν υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία δηλαδή υπάρχει μια περιοχή η οποία συνεχίζεται ε, χορτολεβαδικές εκτάσεις ε, μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας. Δεν διακρίνει κανείς ποιο είναι το σύνορο, αλλά η προστασία είναι διαφορετική και οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται την περιοχή από τις δύο μεριές σύνορων δεν έχουν αντιθεί ποτέ. Οπότε νομίζω καλό θα είναι να σκέφτονται τι γίνεται και στην άλλη μεριά των σύνορων και να προωθήσουμε λίγο περισσότερο την διασυνοριακή συνεργασία κάποια άλλα βασικά σημεία και τελειώνω. Βεβαίως η μεγάλη πρόκληση είναι το πώς θα ενσωματώσουμε την βιοπικιλότητα στις άλλους τομείς της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ίδιο ισχύει και για τη χρηματοδότηση. Έχουμε μια πολύ δύσκολη συζήτηση μετά το 2013 για τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013 και να δούμε βέβαια τι γίνεται με το Life Plus που είναι μία από τις λίγες γραμμές του προπολογισμού που αυξάνεται φέτος οι υπόλοιπε μειώνονται οπότε νομίζω πως ε, εντάξει το Life Plus είναι ένα πολύ μικρό και περιορισμένο κομμάτι οπότε θα πρέπει να θέσουμε περισσότερους στόχους και πιο φιλόδοξους για αυτή την πολιτική και να δούμε πώς θα το χρηματοδοτήσουμε είτε ε, από την πλευρά της γεωργίας είτε από την πλευρά της κλιματικής αλλαγής να χρηματοδοτήσουμε κάποιους ε, στόχους ε, βιοπικιλότητας αυτό το οποίο λέμε δηλαδή με ένα σπάρο δυο τριγώνια. Βέβαια όταν μιλάμε για βιοπικιλότητα καλό είναι να μην σκοτώνουμε τα τριγώνια αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης πρέπει να βελτιώσουμε την γνώση μας γιατί τα στατιστικά δεδομένα είναι πάρα πολύ διαφορετικά, το επίπεδο της γνώσης είναι πάρα πολύ διαφορετικό και πρέπει να βελτιωθεί και αναφέρω και κάποιες διεθνείς πτυχές και ελπίζω στην διάσκεψη της ε, Ναγκόγια να γίνει μια ευρεία συζήτηση και μια μεγάλη αντιπροσωπεία και να μην είναι μια υπόθεση μόνο υπουργών ε, περιβάλλοντος μεταξύ τους. Επίσης να δούμε ποια είναι η δυναμική θέσεων εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν από τη βιοπικιλότητα της οικοϊπηρεσίας, τις πράσινες αυτές δουλειές, οι οποίες είναι δουλειές οι οποίες είναι εδώ και δεν μπορούν να εξαχθούν σε άλλα μέρη του κόσμου, κάτι το οποίο είναι θετικό. Τέλος, η μελέτη αυτή μας λέει πως δεν είναι μόνο θέμα οικολογίας κτλ αλλά και θέμα οικονομικό είναι προς το οικονομικό μας συμφέρον να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε το κόστος το οποίο γίνεται για την ε, αποκατάσταση ε, της βιοπικιλότητας δεν συνυπολογίζεται όταν ορίζονται οι τιμές, κάτι το οποίο πρέπει να, να ε, γίνει. για να δούμε πώς θα υπάρξει βεβαίως και κάποια ίσως αποζημίωση κάποιων ανθρώπων που είχαν κάποιες δραστηριότητες. Οπότε αυτά είναι τα βασικά. Είμαι πεπισμένη πως βεβαίως θα γίνουν κάποιες προσπάθειες να προσθεθούν διάφορες αποχρώσεις και Ελπίζω αυτή η έκθεση, η οποία είναι αρκετά περιορισμένη, να καταφέρει να περιγράψει όλη αυτή την ποικιλία της βιοποικιλότητας. Σας ευχαριστώ, κυρία Τελάνγκε. Για την έκθεσή σας και όταν το διαβάζει κανείς βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ ουσία, αναφέρεστε σε πάρα πολλές πτυχές που σχετίζονται με το θέμα και πιστεύω ότι αποτελεί μια εξαιρετική βάση για να μπορέσουμε να αιτιολογήσουμε την απόφαση που θα χρειαστεί να πάρουμε. Δίνω το λόγο πρώτα στην Κάριν Κάλενμπανκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω σε πολλά σημεία με τον Γιώ Λάινεν. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο Ντελάνγκ διότι νομίζω ότι στο δύσκολο αυτό θέμα ε, έβαλε σε λίγο χώρο και χρόνο πάρα πολλά θέματα ε, και ε, από τη μία πλευρά ναι μεν συμφωνούμε αλλά πρέπει επίσης να επιμείνουμε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις για τα μετρά διότι οι στόχοι που είχαμε βάλει για το 2010 δεν έχουν υλοποιηθεί και θα έπρεπε κάποια στιγμή να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Ε, θα ήθελα λοιπόν αυτά να τα συνδυάσω με άλλους τομείς. Δηλαδή ε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει προστασία που να συνδυάζεται με την ε, πρόσβαση και αυτό για να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος και της φύσεως. Διότι είδαμε ότι άλλοι πολιτικοί δεν καταλαβαίνουν καθόλου ότι χρειάζεται προστασία. Ενώ εδώ βλέπω ότι ναι μεν δεν έχετε περιλάβει όλα τα θέματα αλλά θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την ε, υποδομή ε, και την ε, βιομηχανία διότι θα πρέπει να περιλάβουμε όλους τους περιορισμούς των περιοχών της φύσεως που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συνυπολογιστούν κατά την εκπόνηση των μέτρων. Όσον αφορά τις ε, ε, τροπολογίες, ε, νομίζω ότι στο σημείο 7 δεν θα πρέπει να ικανοποιηθούμε με τους στόχους και να τους εμπλουτίσουμε, διότι ουσιαστικά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε κατά προτεραιότητα ορισμένα θέματα. Αλλά πιστεύω ότι βάσει του περιορισμένου χρόνου που έχουμε δεν πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μέτρα τα οποία θα καθυστερήσουν περαιτέρω τις ενέργειές μας όπως παραδείγματο χάρη την αξιολόγηση της κατάστασης ε, διότι όπου ε, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία ακόμη και αν δεν είναι τελείως ενημερωμένα θα πρέπει αμέσως να προχωρήσουμε στη φάση εφαρμογής εκεί που δεν συμφωνώ με την συνάδελφο είναι στο σημείο 15 όταν ε, λέγεται ότι χαιρετήσει την ευελιξία διότι φοβάμαι ότι η ευελιξία μπορεί να οδηγήσει και σε μια ισοπαίδωση προς τα κάτω. Άρα <clears throat> το να χαιρετίζει κανείς την ευελιξία δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Απλούστατα ε, θα έπρεπε να πούμε ότι χρειάζεται σε ορισμένους τομείς ευελιξία στην εφαρμογή. Ε, αλλά να είμαστε πιο ρεαλιστικοί. Επίσης όσον αφορά την ε, δυνατότητα απασχόλησης. Οι φόβοι που υπάρχουν εδώ τις ε, βιομηχανίες κατά της υπερβολικής προστασίας του περιβάλλοντος και των υπερβολικών μέτρων δεν πρέπει να αποβλέπουν σε ένα περιορισμό των δραστηριών τίτων μας διότι ε, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέων επαγγελμάτων και δηλαδή ε, μπορεί κανείς ε, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις περιφέρειες και όχι σε άλλα μέρη. Ε, είναι μία ένδειξη της περιφερειακής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό το οποίο θα ήθελα επιπλέον είναι εφόσον ε, θα πρέπει να υπάρξει προστασία σε όλους τους ε, τομείς της πολιτικής ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να αναφέρονται όλα τα πράγματα με το όνομά τους διότι εφόσον μιλάμε για τα διαρθρωτικά μέτρα θα πρέπει να μην σκεφτούμε μόνο τη δημιουργία δημιουργία θέσεων που θα οδηγήσουν, ε, ε, ε, που θα, ασχοληθούν με την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, τέλος, σαν Αυστριακή θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να φυγεί επίσης. Κάτι το οποίο διαπιστώνουμε συνέχεια και θα πρέπει να ληφθεί η υπόψη σχετικά με τη συζήτηση για την προστασία του κλίματος ε, είναι ότι δεν ε, πρέπει ε, θα πρέπει θα πρέπει να υπάρξει η βιοπικιλότητα την οποία ναι, επιζητούμε αλλά να μην ε, επιτευχθεί εις βάρος άλλων στοιχείων. Τέλος, όσον αφορά τις ε, τροπολογίες θα επανέλθουμε, αλλά καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την πολύ καλή αρχική εργασία που έχει γίνει και η οποία θα μας επιτρέψει απλώς να προβούμε σε λίγες προσθήκες. Ευχαριστώ, Κάριν Κάλενμπαχ ε, ε, θα πρέπει ίσως να ξεκινάει το ρολόι για να βλέπει ο καθένας πόση ώρα μιλάει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Νομίζω πως αναφέρονται τα σημαντικότερα σημεία, οπότε είναι μια εξαιρετική βάση για να εργαστούμε περαιτέρω. Υπήρχε μια καθυστέρηση, είναι κρίμα που δεν την είχαμε νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, φωνάζω και από ενθουσιασμό βεβαίω, γιατί λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει πράγματι η συγκήτρια είχε περιορισμένο χώρο, οπότε μπορούμε να εργαστούμε. Αυτό το οποίο νομίζω λείπει και είναι σημαντικό και δεν έχει να κάνει με κάποια συγκεκριμένα σημεία, δεν υπάρχει εδώ πέρα ένα αίσθημα του κατεπήγοντος είναι πολύ άσχημη η κατάσταση στην βιοπικιλότητα. Το είδαμε και πριν από δύο εβδομάδες με την έκθεση της UNEP. Είδαμε τι γίνεται με την BP στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ε, την λεωφόρα πέτρα λεωφόρα όμως στον ε, Καναδά, εξακολουθούμε να ζητούν παντού πρωτοσύλλες και κινδυνεύει έτσι η βιοπικιλότητα. Και νομίζω πως θα πρέπει το ψήφισμα αυτό να αντικατοπτρίζει καλύτερα το αίσθημα αυτό του κατεπήγοντος. Αυτό το οποίο επίσης λείπει εδώ πέρα και θα σκεφτώ λίγο τον ε, Bill Clinton ε, είναι αυτό το οποίο είχε πει στον George Bush ότι βεβαίως η οικονομία είναι το, το θέμα. Οπότε εγώ είμαι πεπισμένος πως ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε την βιοπικιλότητα είναι με το να την ενσωματώσουμε στην παγκόσμια οικονομία. Θα αναφέρω κάποια βασικά σημεία. Καταρχήν βεβαίως εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τώρα 2000 και η οδηγία ε, για τα πτηνά και το Habitat. Αυτό το οποίο λείπει όμως είναι το να τονίσουμε τι φοβερή επιτυχία είναι το Natura 2000. Αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει εντός της Ευρώπης με αυτό το έργο προστασίας φύσης είναι φανταστικό. Και θα ήθελα να σας προσκαλέσω επί την ευκαιρία την ερχόμενη Τρίτη σε μια φωτογραφική έκθεση εντός του Κοινοβουλίου ακριβώς για την ομορφιά και την δύναμη της ε, ευρωπαϊκής φύσης. Ε, την άλλη τρίτη έξι ώρα στο Ισόγειο, The Wild Wonders λέγεται η έκθεση. Οπότε, για την ευελιξία, το αναφέρει αρκετές φορές η Κομισιόν, πως υπάρχει αρκετή ευελιξία, πως σε κάποια κράτη-μέλη ε, υπάρχει λιγότερη ευελιξία στην ερμηνεία, αλλά αυτό δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θέμα εθνικής ε, πολιτικής. Έχω μία ερώτηση τώρα για το σημείο 18, το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως, γιατί καλεί την Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο σε οικοστημικές υπηρεσίες και την προσαρμοστικότητα κτλ. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό να αυξηθεί η πίεση στα οικοστήματα. Αντιθέτως πρέπει να μειωθεί η πίεση στα οικοστήματα για να επανέλθουν από μόνα τους. Αλλά νομίζω θα μπορούσε να το εξηγήσει αυτό η συγκεκριτή. Τώρα όσον αφορά την ενσωμάτωση άλλων πολιτικών. Για να είμαι ειλικρινής, ε, αυτό είναι το σημείο κλειδί. Ε, κύριε Πρόεδρε, βλέπω είστε έτοιμος ε, να πατήσετε το κουμπί. Λοιπόν, αυτό είναι το, το κλειδί. δηλαδή, ειδικά οι πολιτικοί της αλλιές και άλλες πολιτικές θα παίξουν κρίσιμο ρόλο πρόσφατα βγήκε και η έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για τις επιπτώσεις που έχει η πολιτική γεωργία στην βιοπικιλότητα και είναι πραγματικά ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες ε, μείωση τη βιοπικιλότητα. Ε, πρέπει να δούμε επίσης την βιομηχανική αλλιευτική πολιτική, μία από τι μεγάλες αδυναμίες Ευρώπης, δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο ε, αδειάζουμε τις θάλασσες από ψάρια θα έπρεπε να ενισχυθεί ίσως κάπου η έκθεση. Τώρα η χρηματοδότηση. Πρέπει να δούμε πιο επικριτικά τις ε, επιδοτήσεις που δίνει η ίδια η Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές επιδοτήσεις που έχουν αρνητική επίπτωση στη βιοπικιλότητα και κατά την άποψή μου μπορούν να καταργηθούν. Όσον αφορά λοιπόν την χρηματοδότηση και τη μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτική. είναι αναγκαίο ο προϋπολογισμός που έχουμε για τη Γεωργία να μειωθεί και να δίνουμε λιγότερα λεφτά στη Γεωργία και να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά για να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα και να αποκαταστήσουμε τη βιοπικιλότητα. Συχνά μάλιστα μιλάμε για τις ίδιες περιοχές όπου τώρα ε, βόσκουν γελάδες. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, το διεθνές κομμάτι ως ε, κοινοβούλιο. έχουμε και ξεχωριστό ψήφισμα για τη διάσκεψη της Ναγκόγια. Θα κινητοποιηθούμε. Νομίζω πως πρέπει να είμαστε πολύ πιο επικριτικοί εναντί τρίτων χωρών. Είμαστε πολύ ελκυστικοί ε, για τις υπόλοιπες χώρες. Είμαστε 500 εκατομμύρια καταναλωτές, καταναλωτές που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτή είναι η μεγάλη οικονομική μας δύναμη την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προτιμήσουμε ε, να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προϊόντα ε, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη βέβαια στην βιοπικιλότητα. Τέλος, πρέπει να πάμε προς την σύσταση ενός διεθνούς πάνελ για την βιοπικιλότητα, κάτι σαν αυτό που έχουμε για το κλίμα γιατί βεβαίως το να μετράμε είναι γνώση. Και δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για τη βιοπικιλότητα. Είναι δύσκολο να βασιστούμε σε ακριβή δεδομένα. Βεβαίως ε, αυτό απασχολεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Περιβάλλοντος, αλλά καλό είναι να έχουμε ένα τέτοιο πάνελ. Θα μείνω σε αυτά αυτή τη στιγμή κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ξέρω πόσο σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό και την άλλη εβδομάδα θα δούμε τον ο, χώρο, ο, της φύσεως. Είναι για τα ζώα ή ταινία. Αλλά αντιλαμβάνουμε ότι είναι ταινία. Ωραία. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή η συνεισφορά είναι άκρος ε, σημαντική. έτσι ώστε να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στους πόρους που θα πρέπει να δοθούν για την βιοπικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντελάνγκ για την εργασία της γιατί μιλά για την καταπολέμηση της απώλειας της βιοπικιλότητας και την ανάγκη του να εντάξουμε τη βιοπικιλότητα σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές. Έτσι μπορεί το Κοινοβούλιο να λάβει θέση και υπέρ της προστασίας της βιοπικιλότητας και να προωθήσει μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική έτσι ώστε η επιβίωση να μην αφορά το θέμα της διατήρησης και ε, ανάπτυξης, αλλά να υπάρχει ανάπτυξη στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό σκέλος. Δηλαδή να προβάλλουμε μια νέα οικονομική στρατηγική. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή σε ορισμένα σημεία, ότι θα πρέπει δηλαδή να δούμε ε, τα οικοσυστήματα, τα ενδιαιτήματα και να βρούμε και τα κατάλληλα οικονομικά μέσα τα οποία θα πρέπει να αυξηθούν. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι όροι που διέπουν αυτό το πλαίσιο. Να μιλήσουμε για αλία, για μεταφορά, για συνοχή και μια γενικότερη συνοχή των πολιτικών μας και να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει οδηγία για τη γη, για τα είδη τα οποία μας κατακλείζουν και για τη χρήση της ξυλίας. Ε, υπάρχει ε, άρρηκτος δεσμός μεταξύ ανθρωπότητας και βιοπικιλότητας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άρρηκτος αυτός δεσμός αφορά το 70% του πληθυσμού της γης που ζει σε αγροτικές περιοχές στο νότιο ημισφαίριο. 1,6 δις ανθρώπων που εξαρτώνται από την ε, δασοκομεία. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράζω τη λύπη μου διότι η στρατηγική 2020 δεν μιλά για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Εάν συμφωνούμε λοιπόν ότι το θέμα είναι κατεπήγον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο σημείο 8 ε, εάν οι οικονομίες μας και η ζωή μας εξαρτάται από την βιοπικιλότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία επιφύλαξη. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μελέτη αντικτύπου πριν να ορίσουμε τους στόχους. Για άλλη μία φορά ευχαριστώ την κυρία Ντελάνγκ για την ποιότητα της έκθεσης θα υποβάλουμε τροπολογίες για να ενισχύσουμε αυτή την πρόταση. Και η Ζούλη Κέρλινγκ. Η Ελίζα Φερέιρα. Ούτε. Είναι η Ευχαριστώ. Και εδώ αντιμετωπίζουμε ένα θέμα το οποίο μας ε, απασχολεί άμεσα. Μιλάμε για την ποιότητα της ζωής, την ανθρώπινη ε, ζωή και όλων των ζωικών ειδών. Όταν συντάσσουμε αυτά τα έγγραφα, πολλές φορές υπερβάλλουμε στην έκφρασή μας ή προβάλλουμε αντιφατικά στοιχεία δηλαδή το γεγονός ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τις απώλειες από την ε, βιοπικιλότητα σημαίνει ότι σταματάμε την εξέλιξη των ειδών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επέλθει καμία αλλαγή. Θα μείνουμε στην εποχή της, ε, του, στη λίθινη εποχή και θα ήμασταν δεινόσαυροι σήμερα βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής, αλλά αν είμαστε σοβαροί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για, για το ότι σταματάμε την εξελικτική πορεία των ειδών, διότι πολλά είδη έχουν εξαφανιστεί και άλλα έχουν ε, γεννηθεί. Γιατί αυτή είναι η ζωή του ε, πλανήτη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανακοπή λοιπόν της πορείας. Επίσης μιλάμε για στοιχεία που λείπουν και μιλάμε για τι στοιχίζει ετησίω η απώλεια βιοπικιλότητα. Μα τα στοιχεία υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Τα στοιχεία υπάρχουν. Γιατί λέτε ότι δεν υπάρχουν. Και η έκθεση έχει έναν αρνητικό χαρακτήρα. Όμως έχουν ε, έχουν ε, γίνει πολλές προσπάθειες από τοπική αυτοδιοίκηση, από τις περιφέρειες και επανεμφανίστηκαν ήδη που είχαν εξαφανιστεί. Παραδείγματος χάρη πολλά αρπακτικά, πολλά ε, πτηνά που ζουν στα ύδατα, πολλά αμφίβια. Ε, τότε τι να κάνουμε, να, κλείσουμε και τη διόρυγα του Σουέζ. Αυτή η, πορεία που λέτε δεν είναι ανελικτική. Μιλάμε για πανίδα και χλωρίδα. Δηλαδή πολλά είδη ε, εξαφανίστηκαν μετά από τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ. Τι να κάνουμε, να την ξανακλείσουμε τη διόρυγα για να εμφανιστούν, επαναεμφανιστούν αυτά τα είδη. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς οι, κλιμα... οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν τη βιοπικιλότητα. Βεβαίως, αν αλλάξουν οι θερμοκρασίες του πλανήτη, η θερμοκρασία του πλανήτη, βεβαίως θα αλλάξουν και τα είδη τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν. οι πολλοί Αφρικανοί ε, βρέθηκαν προς το, τη βορρά, το βορρά της Ευρώπης όταν αποχώρησαν οι πάγοι. Μετά δηλαδή από την εποχή των παγετώνων. Δεν νομίζω ότι εμείς ως ευρωβουλευτές θα ήμασταν πιο ε, δυνατοί όταν θέλουμε να ανασχέσουμε μια απορία. Πιστεύω στην προστασία των ειδών. Μιλάμε για την εναλλακτική επίσης αλία για να μιλήσουμε για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Μην ξεχνάμε ότι η υδατοκαλλιέργεια δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και ζημίες στη βιοπικιλότητα είχαμε, ε, πολύ, είχαμε μια μεγάλη εισβολή ε, ειδών, από τα ε, γλυκά ύδατα που ήρθαν προς τα δικά μας μέρη από την Αμερική. Γιατί ξέρουμε ότι, πολύ καλά ότι η υδατοκαλλιέργεια δεν είναι πανάκια για όλα. Δηλαδή μη μιλάμε και για ασφικτική προστασία. Η κορμοράνη επειδή απαγορεύθηκε το κυνήγι τους έχουν κατακλείσει τη γη. Και άρα σήμερα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που ε, τώρα πια είναι έξω από τις δυνατότητες μας, διότι ένας κορμοράνος τρώει 400 ε, ε, γραμμάρια ε, ψαριών ημερησίως. Υπάρχουν και άλλα είδη, ας πούμε ο ξύριγχος στην Ιταλία, ο οποίος δεν επιτρέπεται να αλλιευθεί. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Λιγουρίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πτηνά τα οποία επειδή ακριβώς δεν μπορούν να κυνηγηθούν, τι κάνουν, μας τρώνε τις ελιές στη Λιγουρία. Άρα όταν γράφουμε την ιστορία να την γράψουμε σωστά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για βιοπικιλότητα, ας μην προβαίνουμε σε ασφικτική εποπτεία και έλεγχο. Äh, äh. Ναι, ε, αυτή είναι μία αντιφατική ε, επιχειρηματολογία η οποία παρουσιάστηκε εδώ. Και ίσως καλό θα ήταν να ξέραμε τι γινόταν την ε, στη λίθινη εποχή. Αλλά ε, βλέπετε ότι ο χρόνος τρέχει και ο Πέτερ Βαντάλεν είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα περάσουμε τώρα στην ε, προϊστορία. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο, στο 2010, το έτος της ε, βιοπικελότητας όπου δυστυχώς βλέπουμε πως η βιοποικιλότητα υποχωρεί. Και είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη ζωή μας, για τη ζωή στη γη, ως βάση του ανθρώπου και των ζώων. Και εγώ εξεπλάγιν ευχάριστα από την ε, έκθεση της συναδέλφου Ντελάνγκε, από το πράσινο χρώμα που διατρέχει την έκθεση. Από την άλλη πλευρά έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξη σε κάποια σημεία. Έχω και ένα συγκεκριμένο ερώτημα επίσης και μία πρόταση. Ας κάνω τώρα την πρόταση. Στην ε, παραγραφό 32 αναφέρει πως ε, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Συμφωνώ, αλλά είναι πολύ φιλική αυτή η, η παράγραφος ε, όσον αφορά την ε, επικουρικότητα. Νομίζω πως ε, πρέπει να δώσουμε μια πιο έντονη όθηση στα κράτη-μέλη. Τέλος αυτό θα γίνει νομίζω με τις τροπολογίες. Το συγκεκριμένο μου ερώτημα τώρα αφορά τις επιλογές όσον αφορά αυτό το οποίο λέει π.χ. στην σελίδα 12 για την επικοινωνία που μπορεί να κάνει η Κομισιόν. Εγώ νομίζω πως θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες εξηγήσει για να... Δεν ξέρω να μας εξηγήσει γιατί ε, τι διαλέγει ακριβώς ε, η συγκέντρα. Νομίζω πως διαλέγει την επιλογή 4 δεν ξέρω. Νομίζω πως θα πρέπει να γράψουμε ξεκάθαρα την επιλογή, την επιλογή 4, εν πάση περιπτώσει, αυτή που προτιμάει η συγκίτρια εντό τη έκθεση. Νομίζω εγώ θα προτείνω μια τροπολογία. Πρέπει να είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το κείμενο εδώ πέρα, γιατί νομίζω πως πραγματικά πρέπει να είναι ρητή η θέση μας εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, σαφή λόγια. Τουλάχιστον Ολλανδικά είναι ε, σαφές ενώ δεν μπορεί να είναι ασαφές τα Ολλανδικά αφού ήταν και η συγγήτρια ε, Ολλανδέζα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πρέπει σε 10 λεπτά να φύγω για την αντιπροσωπή της Παλαιστίνης αλλά υπήρχαν πριν πολλά χρόνια πολύ περισσότερα ψάρια τα οποία ξεφορτωνόντουσαν στην Βρετανία από ό,τι τώρα διότι τώρα όλες οι αλληλίες είναι υποπίεση τα συμφέροντά μας τα αλλιευτικά έχουν μειωθεί πάρα πολύ διότι οι ε, χώρες μας ε, οι θάλασσές μας μπορούν να θρέψουν πολύ περισσότερα ψάρια από αυτά που είναι μέσα αλλά το οικονομικό αυτό πρόγραμμα είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε στους υπουργούς τις μεταρρυθμιστικές προοπτικές αλλά βλέπουμε ότι ε, από την άλλη πλευρά ε, στρέφουμε τα είδη και ε, τα πλάσματα του Θεού πιο γρήγορα από ότι οποιαδήποτε άλλη εποχή από όταν τελείωσε η εποχή των δεινοσαύρων. Τι μπορούμε να αλλάξουμε. Καταρχήν τη νομοθεσία. Μπορούμε να ρυθμίσουμε θέματα μειώνοντας ορισμένα ζύζανιοκτώνα τα οποία σκοτώνουν και τη ζωή. Επίσης ε, ζητώντας από τους ε, γεωργούς να αφήνουν χωρίς να καλλιεργούν ένα μέρος των αγρών τους για να διατηρήσουν τη βιοπικιλότητα. Από την άλλη πλευρά όμως χρησιμοποιούμε και μεθόδους που ορισμένοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν και πετάμε ε, χρήματα ε, για τις βέλτιστες πρακτικές, ε, για τα κίνητρα, τα θετικά ε, για την βιοπικιλότητα αλλά ε, δεν έχουμε και τόσα χρήματα, ε, είναι περιορισμένοι οι πόροι μας. Οπότε αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσουμε να στραφούμε προς εργαλεία της αγοράς για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτές τις αντιφατικές ε, μεθόδους. Διότι βλέπω ότι παραδείγματο χάρη προσπαθούμε να περιορίσουμε ε, την ε, βιομηχανία, να την υποχρεώσουμε να αντιδρά θετικά και η Επίτροπος εχθές είπε ότι θα ήθελε να υπάρχουν εμπορεύσιμες άδειε για τα αλλιευτικά προϊόντα όπου έχουν χρησιμοποιηθεί οδήγησαν αμέσως σε μείωση της υπερβολικής χωρητικότητας και άρα δίδουν ελπίζουμε και περισσότερα χρήματα στους ε, τους <clears throat> Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο εργαλείο της αγοράς το οποίο ίσως είναι ατελές αλλά είναι μια θετική πρόοδος προς τα εμπρός. Και όταν κοιτάξουμε τη γεωργία, όταν κοιτάξουμε τον τεράστιο όγκο του, της γης που μας περιβάλλει αναρωτιέμαι τι μέτρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θα ήθελα κάποιος να μπορεί κάτι να προτείνει τι θα μπορούμε να πτύξουμε, να διερευνήσουμε αλλά τι είναι αυτά ε, έχει μια ιδέα, κάποια ιδέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η συγγήτρια, διότι αν δεν βρούμε κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα της ανθρωπότητος και η δυνατότητα εκμεταλλεύσεως δεν ε, ισοζυγιστούν, νομίζω ότι βαίνουμε προς την καταστροφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να δούμε, θα μας πει μετά η συγγήτρια τι ε, μέτρα σκέφτεται να εφαρμόσει στην αγορά. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια είπε σαφώς ότι οι στόχοι αυτοί για το 2010 δεν μπορούν να υλοποιηθούν και ότι απέχουμε πολύ από τους στόχους αυτούς. Δεν ξέρω εάν έχετε δει το αιτιολογικό σκέλος του εγγράφου όπου υπάρχουν ανησυχητικοί αριθμοί και στοιχεία. Τουλάχιστον εγώ πλάγιν. Και αυτό που διαβάζω εδώ είναι ότι αν η τάση αυτή συνεχίσει τότε μέχρι το 2050 εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα υπάρξει μία μείωση της βιολογικής βιοπικιλότητος ε, για τις πεταλούδες 45% ε, για τα ερπετά επίσης ένα υψηλό ποσοστό δηλαδή υπάρχουν πολλές απώλειες δεν ξέρω πού βρήκε η συγγήτρια αυτά τα στοιχεία εγώ τουλάχιστον δεν τα γνώριζα αλλά εάν ο κίνδυνος όντως είναι τόσο μεγάλο το 2050 είναι μόνο μια μισή γενιά μπροστά. Δηλαδή ε, το παιδί μου θα έχει τότε την ηλικία, το νεότερο παιδί μου. Άρα θα ζήσει την εποχή εκείνη. Οπότε δεν εύχομαι να υπάρχει μία τέτοια ζωή όπου θα ισχύσουν αυτές οι προϋποθέσεις. Αυτό όμως το οποίο σκέφτομαι είναι ότι υπάρχουν και λήψεις στην έκθεση αυτή και θα παρακαλούσα την εισηγήτρια να συμπληρώσει αυτό το έγγραφο, διότι δεν ξέρουμε παραδείγματο χάρη ποιοι είναι οι στόχοι, γιατί δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, γιατί απέχουμε τόσο πολύ από την επίτευξη των ε, στόχων μας, δηλαδή ποιο είναι το παρασκήνιο και μπορώ απλώς να ερωτώ, δεν γνωρίζω τις απαντήσεις της ερωτήσεις μου. Η υποδομή των μεταφορών παραδείγματο χάρη, μήπως και αυτή έχει μείνει πίσω, μήπως αυτό, σε αυτό οφείλεται ότι μειώνεται η βιολογική βιοπικιλότης, διότι οι περιοχές της Natura 2000 επίσης αναφέρονται, αλλά βλέπουμε ότι στις περιοχές αυτές ε, διέρχονται ε, αυτοκινητόδρομοι. Επίσης οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία γνωρίζουμε πώς λειτουργούν αλλά υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε κατά τρόπο ώστε ε, να μειώσουμε τους κινδύνους οι οποίοι δημιουργούνται στην απασχόληση. Ε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει κάποιο ρόλο για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχει σχέση με τους μηχανισμούς αποφάσεως, διότι έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρει αριστερά τι πει ή δεξιά. Παραδείγματος ε, χάρη, τη Δευτέρα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ε, οδικό δίκτυο, την Τρίτη βλέπουμε όμως ότι ε, πολλαπλασιάζονται ε, διάφορα στοιχεία. Την Τετάρτη θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Δούναβη, αλλά την Πέμπτη πιστεύουμε ότι στην ε, περιοχή εκείνη θα υπάρξει σοβαρή βλάβη. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε πολλές φορές ποιες είναι οι επιπτώσεις των πράξεών μας και δεν ξέρω αν οι στόχοι που αναφέρονται ε, μέσα στο έγγραφο αυτό είναι απλώς ένα ευχολόγιο στο οποίο προσβλέπουμε. Ευχαριστώ. Ε, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει μία συνεκτική πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Κορίν Λεπάζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή για την εκθεσή του που τονίζει ορισμένες δυσκολίες και θα ήθελα να εκφράσω και την ανησυχία μου όταν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο κινείται αυτή η στρατηγική που θα που μας οδηγήσει σε μια γενικότερη ε, πολιτική και αιτιώδη συνάφεια Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους ε, για τους ίδιους λόγους. Εάν μπορούμε να διατηρήσουμε την βιοπικιλότητα, σημαίνει ότι κάναμε τις ε, σωστές επενδύσεις. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μία σωστή αποτίμηση. Ο συνάδελφος είπε ότι είναι αντιφατική πολλές φορές η στόχη μας διότι το θέμα της βιοπικιλότητας δεν είναι οικονομικό αποκλειστικά. Αν λοιπόν δεν το έχουμε ενσωματώσει στους στόχους μας, σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μία νέα προσπάθεια έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε το συλλογικό κόστος και στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να βαστούμε στην έκθεση Stern και ίσως θα πρέπει να τονίσουμε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το συλλογικό κληροδότημα, αυτή τη συλλογική κληρονομιά. Μα υπάρχει έκθεση Στέρν που μιλά για τις οικονομικές ζημίες, απώλειες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ε, απώλεια στη βιοπικιλότητα. Και αυτό δεν το λέει μόνο η έκθεση στερν. Ο Βιτόριο Πρόντι. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ το συνάδελφο για αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να καταδείξουμε ταπεινότητα απέναντι στη φύση και την ανάγκη να μάθουμε περισσότερα για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και στο θέμα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε λεπτομεριακά, ιδιαίτερα σε σχέση με τα τροπικά δάση, μέσα από τα οποία περνάνε ε, ποτάμια που παρουσιάζουν μεγάλη βιοπικιλότητα. Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε απόλυτα το θέμα της ε, βιοπικιλότητας, έτσι ώστε να μιλάμε για μια πραγματική διατήρηση. Μιλάμε για, τις, για την αρχή της προφύλαξης, αλλά δεν γνωρίζουμε επαρκώς την βιοπικιλότητα και όλων αυτών των οικοσυστημάτων για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε. Και βεβαίως ε, πολλές φορές ε, ίσως υπάρχει ε, μία προληπτική δραστηριότητα την οποία θα μπορούσαμε να προωθήσουμε. Έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να αποτιμήσουμε τους αντικτύπους. Το θέμα είναι πολιτισμικό λοιπόν. Να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να αναζητήσουμε τους αντικτύπους της δράσης μας στην, ε, στο περιβάλλον για να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχουν ε, ε, θέματα τα οποία είναι αναπόδραστα. Σε σχέση ας πούμε με το ωμέγα 3 και ωμέγα 6, αυτά τα ιχνοστοιχεία. Το ωμέγα 3 μας το δίνουν τα ψάρια. Εάν έχουμε λιγότερα ε, αλλιευτικά είδη, αυτό θα έχει επιπτώσει στον άνθρωπο και στην ευφία μας, στους ανθρώπους και στην ευφία τους, διότι τα λιπαρά ω 3 είναι απολύτως απαραίτητα για τον άνθρωπο για το νευρικό του σύστημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά και θα πρέπει να αναζητήσουμε την ελαχιστοποίηση ε, των επιπτώσεων της ε, ανθρώπινης δραστηριότητας. Ας μιλήσουμε και για την ανθρώπινη οικολογία. Στα Ηνωμένα Έθνη, κατά τα τέλη Απριλίου, έλαβε χώρα το μόνιμο πάνελ που ασχολήθηκε με τους αυτόχθονες πληθυσμούς της γης και βλέπουμε ότι πολλοί, πολλοί αυτόχθονες πληθυσμοί αρχίζουν να εκλείπουν και αυτό έχει σχέση με την βία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να δείξει ότι πρέπει να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση προς τους συνανθρώπους μας. Μάλιστα μάθαμε κάποια πράγματα, το ω3 είναι καλό για την νοημοσύνη, οπότε ποιο τρώει ψάρια είναι πιο έξυπνος. Ισχύει και για τα ψάρια, για το κρέας αυτό ή μόνο για το ψάρι. Α, για το ψάρι. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω τη μητρική μου καθώς είναι η ίδια με τις συγκεκριές. Κυρία συγκήτρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση αυτή και έχει πάρα πολύ καλές ε, πτυχές ε, μέσα. Βεβαίως ε, δεν είμαι και τελείως ικανοποιημένος. Θα ήθελα να σας πω πως αυτό το οποίο λείπει είναι η φιλοδοξία για το μέλλον. Γιατί ξεκινάτε καλά και λέτε πως έχουμε προβλήματα και δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα, άρα ότι δεν κάνουμε αρκετά ως Ευρώπη. Και μετά λέτε τι θα γίνει με το Natura 2000, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Πώς θα έχουμε επιτύχει τους στόχους του 2020. Αυτό μου λείπει από την έκθεση. Δεν πετυχαίνουμε τους στόχους τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε τελείως διαφορετικά λοιπόν για να τους επιτύχουμε στο μέλλον. Αυτή η φιλοδοξία μου λείπει. Γιατί μπορούμε νομίζω να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αυτή λοιπόν η φιλοδοξία για το μέλλον πρέπει να υπάρχει και θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι θα γίνει με την πολιτική της γεωργίας, ο προϋπολογισμός αυτός να δώσει κάποια λεφτά και για υπηρεσίες οικοσυστήματος και να δούμε το τι θα γίνει με την αηφόρο γεωργία λέτε σε ευαίσθητες περιοχές. Όχι, τέλος. Αηφόρος γεωργία, τέλος. Όλη η γεωργία να γίνει αηφόρος. Επίσης, λέτε αηφόρος, ε, να δούμε την το καλλιέργεια. Όχι. Πρέπει να πάμε στην αηφόρο καλλιέργεια. τελεία. Γιατί είναι πολύ προσεκτικές εδώ πέρα οι διατύπωσες σας. Θέμε πραγματικά μία γνήσια αλλαγή εάν είναι πράγματι να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα. Τέλος, πρέπει να υπάρχει συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής και με τη Γεωργία και με το Ταμείο Συνοχής climate proofing που λέμε και πρέπει να υπάρχει και biodiversity proofing, να υπάρχει και μια θωράκιση από πλευράς βιοπικιλότητας, αλλιώς να μην γίνονται τα έργα. Αυτά λοιπόν από αυτή την έκθεση και αυτό το οποίο θα θέλουμε βεβαίω. Έχουμε κριτήρια εφορία για τα βιοκαύσιμα, αλλά για την βιοενέργεια γενικότερα δεν ε, έχει κάνει τίποτα η Λέει θα το κάνουμε, αλλά το χρειαζόμαστε αυτό για κάθε χρήση γης, για παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες που θέμε να δούμε στην έκθεση ε, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας το 2020 για να είναι ικανοποιημένη και η συγκέντρια και να μπορέσουμε να πούμε τότε πως επιτέλους καταφέρουμε κάτι και δεν βάλαμε μόνο στόχους. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δείξω τρία θέματα. Θα πρέπει αυτή η έκθεση και να ευχαριστήσω βεβαίως ε, το συντάκτη. Είναι ένα πρώτο βήμα για να προωθήσουμε περισσότερο το θέμα της πρόληψης των ε, καταστροφών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την ε, εισηγήτρια, διότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας. Η Κορίν Λεπάζ μας ε, μίλησε για τις ε, καταστροφές στην Ευρώπη και υπερασπίστηκε και τα θύματα αυτών των καταστροφών. Ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει στις ακτές της Αμερικής τι έγινε από την, από την BP, πώς κατέστρεψε η BP τη βιοπικιλότητα που θα έχει αναρρύθμιτες επιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν, όπως είπε η Κορίν Λεπάς, να τονίσουμε ότι θα πρέπει να προβάλλουμε μία πολιτική πρόληψης. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε πολλούς ποταμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον οποίο η κατάσταση επιδεινούται. Αυτό το βλέπετε είτε σαν ε, τουρίστες, είτε σαν ε, επισκέπτες στο Παρίσι. Μην πάτε στο Σικουάνα να ψαρέψετε ή να φάτε ψάρια από το Σικουάνα. Το Πυριλένιο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες τα ψάρια του Σικουάνα και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και οι ενδυνάμοι καταναλωτές θα αντιμετώπισαν μεγάλους κινδύνους. Άρα θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις σε σχέση με την ποιότητα των υδάτων και των ποταμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε αυτά που είπατε πριν, ως προς την διασυνοριακή συνεργασία, Νομίζω ότι και εδώ στην έκθεσή σας θα πρέπει να παρακινήσουμε την χρηματοδότηση, τη σημαντική ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, διασυνοριακή συνεργασία με την, ε, με την Μαρτίνο Μπρί. Συνεργαζόμαστε μεταξύ Βαλωνίας, Φλάνδρας και Γαλλίας ε, για δύο εκατομμύρια κατοίκους και το πρώτο πρόγραμμα ε, διετές σχετίζεται με την ανάπτυξη της ε, βιοπικιλότητας. Αν μπορούμε λοιπόν να έχουμε και μία χρηματοδοτική παρακίνηση, ας το πω, αυτό, ας το πω έτσι, για τη διασυνοριακή συνεργασία, θα ήταν ένα σωστό βήμα προς την καλή κατεύθυνση. Δεν θα ψαρέψουμε στο Σικουάνα. Κάποια στιγμή όμως θέλουμε να ψαρεύουμε και στο Σικουάνα και να τρώμε τα ψάρια του. Ε, η Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μια καλή έκθεση της Έστερ Ντελάνιε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να διατηρήσουμε και να σεβαστούμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, σχετικά με τη βιοπικιλότητα. Και εδώ έχουμε ένα σενάριο καταστροφικό κοσμογονίας. Βλέπω ότι ορισμένοι λείπτουν, ενώ βλέπουμε ότι ε, η πέθρος ανθίζει ακόμη και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την φύση. Ζούμε σε μια θαυμάσια περιοχή, ε, διατηρούμε τη φύση αυτή και γι' αυτό ε, αναφέρομαι στη γεωργία που όλα αυτά μας τα εγγυάται διότι στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική λέγεται τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι γεωργοί. Δηλαδή όλοι οι ευρωπαϊκοί πόροι ε, γίνονται μόνο εφόσον ε, υπάρχει ε, πολλαπλή συμμόρφωση και βλέπουμε ότι υπάρχουν θεσμοθετημένα μέτρα με τις οδηγίες που επιτρέπουν να προχωράμε σωστά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό και των καλών σημείων. Ε, τι έγινε με τα φυτοφάρμακα διότι τώρα ε, έχουμε ορισμένα ζυζάνια τα οποία όμως ε, προστατεύουν ορισμένα θέματα και όλα αυτά εξασφαλίζει ότι υπάρχει βιοπικιλότης. Άρα πρέπει να τονίζουμε και τα θετικά στοιχεία και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν προς της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η Natura ομάδες πάντοτε ε, μπορεί να κατηγορείται. Συμφωνώ με την Κορίν Λεπάζο ότι πρέπει να κάνουμε μία μελέτη κόστους και αποτελέσματος σχετικά με τη βιοπικιλότητα και δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα η ομίγυρης εδώ διότι ξέρω στην περιοχή μου θέλουμε να κάνουμε έναν δρόμο και όλοι φέρνουν προσκόμματα και το κόστος έχει διονγκωθεί πάρα πολύ. Ο πρόεδρος ξέρει γιατί ομιλώ. Θα έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την καλή βάση της εκθέσεως Ντελάνιε για μία έκθεση για την προστασία του εδάφους. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε και πρέπει να τονιστεί. Δηλαδή αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει πρέπει να αναφέρονται με το όνομά τους. Πρόκειται για μία καλή έκθεση αυτή η έκθεση Ντελάνιε και θα έπρεπε να τη στηρίξουμε και στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εάν ε, η ε, γεωργία είναι πάντοτε τόσο ποικίλη όπως ε, στην κοιλάδα του ποταμού Μοζέλα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αλλά δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω μόνο μερικά λόγια. Δηλαδή, Εκτιμώ ιδιαίτερο την έκθεση αυτή και ιδίω διότι είναι πολύ δυσάρεστο για μένα να ακούω ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία παραμένει στο επίπεδο της ε, προσπα... Ε, προστασίας των ειδών και όχι βιοπικιλότητας. Το Natura 2000 δεν προστατεύει την βιοπικιλότητα αλλά τα είδη ενώ εμείς θέλουμε να καλύψουμε ε, όλο το, φάσμα. Ευχαριστώ. 20 είχαν ζητήσει το λόγο. Βλέπετε δηλαδή ότι το θέμα της βιοπικιλότητος είναι κάτι το οποίο να απασχολεί πολλούς και τώρα η συγγήτρια μπορεί να απαντήσει στη σειρά των παρατηρήσεων που έγιναν. Ο συνάδελφος Ρώση που δεν είναι πια εδώ μας είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί ανέφερθηκε στους κορμοράνους ε, παραδείγματος χάρη που πλέον δεν, δεν έχουν μια ε, ισοσκελισμένη ύπαρξη και θέλουμε να προστατεύσουμε όλα τα είδη όλα αυτά είναι ε, μέρος της προστασίας της φύσεως διότι η φύση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ε, βρίσκει πάντοτε κάποια άλλη ισορροπία αλλά στο δικό μας τομέα ίσως η έκβαση είναι αρνητική. Άρα η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα τα οποία τέθησαν απευθεία σε μένα. Ξεκινήσω με την κυρία Κάντεμπαχ. Ε, ήταν καλές οι προτάσεις της για τροπολογίες. Ευχαρίστως να συμπεριληφθούν τομείς όπως οι μεταφορές, υποδομές, ε, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο πράγματι γιατί είναι καλά τα παραδείγματα. Συμφωνώ πράγματι. Νομίζω βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Το σημείο 7 τώρα που λέτε την αύξηση της απώλειας, ε, ναι δεν αρκεί γιατί στο σημείο 8 και στο 9 αναφέρω πολύ συγκεκριμένα την αποκατάσταση και το τι γίνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Οπότε απαντάμε αμέσως και στο ερώτημα Φαντάλιν. Χαίρομαι για το ότι έχουμε τόσους Ολλανδούς συναδέλφους. Φαίνεται πώς πλησιάζουν οι εκλογές στην ε, Ολλανδία. Αλλά να απαντήσω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριο Φαντάλε. Ποιο σενάριο θέμε από τι επιλογέ που έχουμε, που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Ναι, βεβαίω το σενάριο 4. Αν δείτε το 8 και το 9, προφανώ είναι το 4. Δεν είχα αρκετό χώρο για να γράψω, να εξηγήσω πως για εμένα είναι σημαντικός ε, η αξιολόγηση αντικτύπου. Το είπανε πάρα πολύ αυτό και πράγματι σωστή είναι η πρόταση να πούμε πως η αξιολόγηση αντικτύπου δεν είναι δικαιολογία για να μην κάνουμε ε, τίποτα. Αλλά ειδικά εκεί όπου δεν υπάρχουν αριθμοί, γιατί σε άλλα σημεία υπάρχουν αριθμοί, είναι μια νομιμοποίηση για να, γίνει, για να έχουν κάποιο νόημα αυτέ οι συζητήσεις. Γιατί όταν λέμε πως ε, εκεί πέρα δεν ε, είχαμε στοιχεία, δεν είναι αυτό κάποια δικαιολογία. Πράγματι είναι θεμητό νομίζω γιατί συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν είναι να κάνουμε νέες προτάσεις ζητάει νέα στοιχεία. Οπότε νομίζω πως θα βρούμε κάποιον συμβιβασμό. Ο κύριος Χερμπράντι πράγματι ε, λέει πως δεν υπάρχει εδώ πέρα το στοιχείο του κατεπήγοντος Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τέτοια μέσα στην έκθεση. Θα προσπαθήσω να ενσωματώσω την, την πρότασή του. Τώρα μου είπε για το σημείο 18 και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Τι εννοούσαμε εδώ πέρα. Αυτή ήταν η παρατήρηση του συναδέλφου Πότς που λέει πως το Natura 2000 έχει στόχο την προστασία ειδών και πρέπει να περάσουμε στα οικοσυστήματα. Περνάμε λοιπόν να περάσουμε στην διαχείριση ε, περιοχών και βεβαίως το σημείο 18 έχει νόημα να πει να δούμε αυτή την ευρύτερη προσέγγιση. Γι' αυτό μιλάμε για υπηρεσίες οικοσυστημάτων, όχι να πιέσουμε περισσότερο τα οικοσυστήματα, αλλά να δούμε πώς θα αντιδράσουν αυτά υποπίεση. Εάν δείτε, αν σας ενοχλεί αυτή η πρόταση ενδιάμεση να τη βγάλω, αλλά ε, εκεί πέρα το σημείο, η πρόταση αυτή δεν ξεκινάει με το και ιδιαίτερα. Λέει, προτρέπει την Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο σε οικοστημικέ υπηρεσίε και οικοστήματα με ευρία έννοια. Τώρα λείπουν εδώ πέρα κάποια σημεία που ανέφεραν αρκετοί ομιλητές. Δυστυχώς ο κύριος Ρώση έφυγε. Είναι κρίμα ένα τόσο σοβαρό ε, αντικείμενο να να το βλέπουμε. Έτσι λέει πως δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ε, απώλεια. Εγώ μιλάω στην έκθεσή μου για ε, βιοπικιλότητα την οποία προκαλεί ο άνθρωπος, όχι γενικά για την απώλεια βιοπικιλότητας. Δεν μιλάμε για τους ε, δεινόσαυρους και τα λοιπά. αφήσουμε κατά μέρος. Επίσης για τις παρατηρήσεις του για την ηθιοκαλλιέργεια. Ναι, αλλά μιλάμε για αηφόρο η θεοκαλλιέργεια Και εδώ πέρα νομίζω πως μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά νομίζω σωστό είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ντερόση για τα συγκρουόμενα συμφέροντα, γιατί πράγματι προστατεύουμε το ένα είδος και μετά αυτομάτως αναπτύσσεται το άλλο ή απειλείται ένα άλλο. Έχουμε αυτή τη συζήτηση και στην Ολλανδία, γιατί υπάρχουν αυτοί που λένε πως Εάν ε, προστατεύσουμε το ένα είδο πρέπει να διαχειριστούμε και το άλλο. Εάν επιτρέπεται ή όχι κάτι τέτοιο θα δούμε τώρα θα μας πει και η Κομισιόν. Μετά άλλη μια ερώτηση του κυρίου Φαντάλε. Πράγματι πλησιάζουν εκλογές για το σημείο 32 και το τι θα γίνει με τα διορθωτικά ταμεία και τα κονδύλια της ανάπτυξης υπαίθρου. Και το Αγροτικής Ανάπτυξης. Εάν δείτε τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν το τι κάνουν οι χώρες δηλαδή με την δυνατότητα προώθησης της ε, βιοπικιλότητας ε, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές στα ποσοστά αυτά. Π.χ. θα μπορούσαμε να έχουμε μια υποχρεωτική χρήση ενός ελάχιστου ποσοστού από το τα, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Ευχαρίστω να δω αυτή την πρόταση, είναι ενδιαφέρουσα. Επίσης ε, παρατηρήσεις, ε, ναι αυτό το οποίο είπατε για το biodiversity proofing για να είναι θωρακισμένες και από πλευρά βιοπικιλότητας διάφορες πολιτικές και αυτό να το δούμε και θα μείνω σε, σε αυτά. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, οι άμεσες ερωτήσεις προς τα εμένα, τα υπόλοιπα θα τα δούμε αν θα μπορέσουμε νομίζω να συνεργαστούμε για να συμπληρώσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Στο κυρία Ντελάνι. Πολλές φορές εθνικά είμαστε ε, αντιμέτωποι ε, αντίπαλοι, αλλά ευρωπαϊκά είμαστε αλληλέγγυοι και νομίζω ότι αυτό διεφάνηκε στην ομιλία σας παρόλο και αν στη χώρα σας ίσως ε, έχετε μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική σε ένας ακρογωνιαίος λίθος της εργασίας μας και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Καταρχήν η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι μέχρι τις 9 Ιουνίου. Θα ψηφιστεί εδώ ε, στην Επιτροπή 14 Ιουλίου και ε, στην Ολομέλεια θα πάει αργότερα. Ε, και τώρα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Jacqueline Μαγκλέιντ, γνωστή εκτελεστική διευθύντρια της, ε, του Γραφείου Περιβάλλοντος. Ε, μας συγχωρείτε που περιμένατε τόση ώρα. Νομίζαμε θα τελειώσουμε το προηγούμενο σημείο πριν, αλλά είναι σημαντικό ότι ακούσατε γιατί η βιοπικιλότηση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, ο ίδιος όσον αφορά τη διεθνή στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας σας για το 2011. Σήμερα το πρωί η τηλεόραση με ρώτησε τι σημαίνει ε, το EA ε, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και σημαίνει πολλά και έτσι προσλέπουμε στην παρουσίαση την οποία θα κάνετε. Ευχαριστώ θα, θα ήθελα καταρχήν να παρουσιάσω ορισμένα θέματα τα οποία είναι βασικά για τους επόμενους μήνες και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Καταρχήν η, η έκθεση καταγραφής των αερίων του θερμοκηπίου ολοκληρώνεται και θα παρουσιαστεί ε, θα αναφερθώ στο τι έγινε στην πράσινη εβδομάδα για την βιοπικιλότητα και η συζήτηση που ακούσαμε ήταν πολύ σημαντική και μπορούμε να ακούσουμε ε, και να δώσουμε απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα που έθεσαν ε, παριστάμενοι και πέραν αυτού ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την έκθεση προοπτικών που θα παρουσιαστεί στο τέλος του 2010 και θα επανέλθουμε στο το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 διότι οι προτεραιότητές μας αρχίσουν να διασυνδέονται με αυτές των κρατών μελών και τις δικές σας. Όσον αφορά τα ε, αέρια του θερμοκηπίου, ε, Ποιο είναι το μήνυμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το 2008 ξεκίνησε, ε, μειώθηκαν ε, αυτές οι εκπομπές και φτάνουμε εις, ε, το, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή κατά 11,3 χαμηλότερο από το 1990. Αλλά είναι προφανές ότι η ύφεση η οποία ξεκίνησε στο δεύτερο ήμιση του 2008 ε, επηρέασε τη βελτίωση και ιδίως τον τρόπο με τον οποίο παράγονται αυτές οι εκπομπές και επηρέασε την, τις κατασκευές, τις οικοδομές και τις οδικές μεταφορές. Βεβαίως δημιούργησε και μεγαλύτερες μειώσεις το 2009. Άλλωστε οι υψηλέ τιμές άνθρακα και ε, ε, διοξιδίου του άνθρακος ε, ενθάρρυναν τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν πιο καθαρές πηγές ενεργείας αλλά ε, αντιλαμβανόμαστε ότι θα χρειαστούν βασικές αλλαγές στην οικονομία. Ε, υπάρχει επιρροή και βλέπουμε ότι το πρόγραμμα εμπορίας των εκπομπών μειώθηκε κατά 3% πέρυσι. Οπότε όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά αλλά δεν ε, πρέπει να μειώνουμε τις προσπάθειές μας και γι' αυτό θα θέλαμε να υποφεληθούμε αυτή της ευκαιρία για να αυξηθούν οι επενδύσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να υπάρχει μια οικονομία που να χρησιμοποιεί καλύτερα τους πόρους. Όσον αφορά την βιοπικιλότητα, νομίζω ότι αρχίσουμε να καλύπτουμε τα κενά γνώσεων που είχαμε, διότι στις τελευταίες εβδομάδες αντιληφθήκαμε την ανάγκη αναθεωρήσεως και της ε, εκπονήσεως μιας νέας πολιτικής για να μπορέσουμε ε, να ε, καλύψουμε τους στόχους της βιοπικιλότητας μετά το 2010. Άρα αυτό το οποίο κάναμε είναι να καταρτήσουμε μία baseline, μία γραμμή βάσεως που περιλαμβάνονται όχι μόνο τα στοιχεία από τις οδηγίες που έχουμε αλλά που εξετάζει την επιρροή της Ευρώπης διεθνώς και εξετάζει και άλλους τομείς, δηλαδή αλλαγές στη χρήση υγιής, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την αλληλεία, την δασοκομεία και μέσως μας λύνει και ορισμένα θέματα για το μέλλον. Άρα βλέπετε στον πίνακα ότι υπάρχει μία διαφορετική προσέγγιση προσέγγιση. Δηλαδή δεν έχουμε επαρκείς γνώσης αλλά αυτές που έχουμε φτάνουν για να δράσουμε και ε, ε, μόνο 17% του χώρου κατοικίας μας είναι σε καλή κατάσταση. Ένα μεγάλο ποσοστό των ειδών κινδυνεύει με εξαφάνιση και όλα αυτά διότι δεν υπάρχει επαρκής επαγρύπνηση και χρειάζονται περισσότερες πηγές πληροφοριών. Γνωρίζουμε όμως ποια είναι τα κρίσιμα σημεία. Θέλουμε να στηρίξουμε και τη δικιά σας εργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύστημα πληροφοριών στην Ευρώπη που πρέπει να προωθηθεί και για να συνεργαστούμε καλύτερα με ομάδες εθελοντών για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την βιοπικιλότητα και να αποφύγουμε την μείωσή της. Θα είμαι λοιπόν ευτυχής να ακούσω και να απαντήσω σε ερωτήσεις για τη βιοπικιλότητα διότι ε, θέλω να σχολιάσω στη συνέχεια τις ερωτήσεις που ετέθησαν για τους κορμοράνους και για άλλα. Ε, σχετικά με την έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος ξέρετε ότι κάθε πέντε χρόνια καταρτίζουμε μία τέτοια έκθεση και αλλά φέτος το προσεγγίσαμε διαφορετικά εξετάσαμε τα θέματα του περιβάλλοντος αλλά και τις οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις τις επιπτώσεις στην Ευρώπη και ε, ε, ε, τους στόχους αξιολογήσεως. Δηλαδή αν πάμε σωστά, για ποιο λόγο δεν πάμε σωστά και τι πρέπει να γίνει για να διορθωθούν τα σημεία αυτά. Έχουμε κάνει 38 αξιολογήσεις χωρών, έχουμε μία μακροπρόθεσμη διερευνητική αξιολόγηση σε βασικές τάσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον της Ευρώπης και τέλος καταρτίζουμε κάνουμε μία συνθετική έκθεση και το Νοέμβριο μας επιβεβαίωσε ευγενός ο πρόεδρος Μπούζεκ του Ευρωκοινοβουλίου ότι θα παρουσιάσει αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στις 30 Νοεμβρίου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να είσαστε μαζί μας εκείνη την ημέρα και να συμμετάσχετε στο εργαστήριο με ευρωβουλευτές από άλλες επιτροπές επίσης. Δηλαδή φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσω ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το πού βρίσκονται οι προτεραιότητές μας για το μέλλον. Και έρχομαι στο τελευταίο θέμα που είναι το πρόγραμμα εργασίας 2011 για το γραφείο. Διότι έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα που σε δύο εβδομάδες θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι εσείς ακούτε τις πρώτες δηλώσεις μου. Αλλά ουσιαστικά μετά από την παρουσίαση θα υπάρχουν ε, η ουσιαστική επεξεργασία και προσβλέπουμε ε, στο ότι τα άτομα θα εξετάσουν το, την έκθεση αυτή, θα μας πούν τη γνώμη τους και θα δώσουμε και τρία επιπλέον κίνητρα για να συμμετάσχετε σε αυτήν την αλληλεπίδραση. Καταρχήν θα εξετάσουμε κατά μέτωπον την αποτελεσματικότητα των πόρων, την πράσινη οικονομία και ε, το λογιστική του φυσικού οικοσυστήματος, ιδίως σε θέματα της αναλύσεως του κύκλου ζωής, εξετάζοντας την ευρύτερη εικόνα ε, σύμφωνα, που δείχνει πώς έχει κινηθεί ε, η βιομηχανία και η κοινωνία στο παρελθόν. Διότι δεν έχει λόγο να υπάρξει μία ορθολογιστική χρήση ε, μίας πηγής ενεργείας εάν, είσαστε, εάν αποτυχαίνετε στη χρήση άλλων πηγών παραδείγματος χάρη και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με εσάς πιστεύουμε ότι μπορούμε να διευκρινίσουμε τομείς πολιτικής οι οποίοι αν χρησιμοποιηθούν καλύτερα θα μπορέσουν να συμβάλλουν εις την αποτελεσματικότητα δηλαδή συσκευασία των αποβλήτων ε, σπάνια στοιχεία για την ηλεκτρονική βιομηχανία και το καθεξής. Επίσης πιστεύουμε ότι μπορούμε μπορούμε να σας τη γυρίξουμε στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος ε, κατά τρόπον ώστε ε, να ε, μας βοηθήσετε να προωθήσουμε ορισμένα θέματα και πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα διαστήματος θα μπορέσει να συνδυαστεί καλύτερα με τα προγράμματά μας διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μεγάλο ποσοστό δαπανών για το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα πρέπει να δεσμευτεί στον δικό μας τομέα κατά τρόπον ώστε να ε, έχετε τις αναγκαίες αποδείξεις για να καταρτήσετε ε, ασφαλείς και ισχυρές πολιτικές. Και τέλος βλέπουμε ότι είναι κρίσιμο για την Ευρώπη να δείξει τον καλύτερο σε αυτό από πλευράς ευθύνη ε, ε, και από πλευράς πόρων και τέλος να δούμε πόσο συνεργαζόμαστε με τους γειτονές μας διότι ε, ανατολικά και νότια έχουμε καταρτήσει προσπάθειες που πρέπει να ενταθούν ώστε τα διασυνοριακά προβλήματα να λύνονται καλύτερα και να υπάρχει καλύτερη ροή πληροφοριών. Με τη Γενική Διεύθυνση Ρέλεξ και άλλες προσπαθούμε να αναπτύξουμε ε, τις ε, ικανότητες που υπάρχουν, να ε, βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, την βιοποικιλότητα και ούτω καθεξής. Έχοντας μιλήσει με τον κύριο Γκεράντι, μπορώ να σας πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε το πρόγραμμά μας εργασίας και ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει και η δημοσιονομική αρχή. Εσείς όμως πρέπει να μας πείτε αν είμαστε στο σωστό δρόμο και αν υπάρχουν στοιχεία μέσα σε αυτό το σύνολο τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν το νομοθετικό σας πρόγραμμα, αυτό το οποίο έχετε καταρτήσει ή που σκοπεύετε να εκπονήσετε του χρόνου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναφέρετε αρκετά σημαντικά ζητήματα και οπωσδήποτε συνάδελφοι θέλουν να σχολιάσουν. Αναφέρεται ο κ. Βελμπάνη, ο οποίος είναι ο πρώτο ο οποίο θέλει να προσθέσει, βλέπω, νέε ναι, ιδέε και έχει τον λόγο. Um, Θα περιοριστώ κάπως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ζακλίν Μακλέιτ που βρίσκεται εδώ μεταξύ μα Είναι πολύ καλό να έρχεστε εδώ από καιρού εις για να ε, μοιραζόμαστε τις ε, γνώσεις μας. Είχα την τιμή να έρθω σε επαφή με τον οργανισμό σας. Ε, επισκεφτήκαμε το Φεβρουάριο στην Κοπενχάγη και θα πρέπει να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο επαγγελματισμός που σας διακατέχει θα ήθελα να παροτρύνω όλα τα μέλη να κάνουν το ίδιο, να σας επισκεφτούμε δηλαδή. Ε, ως επίσημη αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχω ένα ερώτημα σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Βεβαίως ε, έχουν μειωθεί και ε, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης εσείς είπατε ότι δεν είναι μόνο θέμα ύφεση, είναι και οι διαρθρωτικές αλλαγές. Θα ήθελα να ακούσω ε, ορισμένες από αυτές. Εξαιτίας λοιπόν της ύφεση δαπανίσαμε λιγότερα χρήματα στην ε, καινοτομία εξαιτίας αυτής της ε, τάσης, γιατί νομίζουμε ότι κάνουμε το σωστό. Θα δούμε πότε θα ανακάμψει η οικονομία εκ νέου, αλλά βρισκόμαστε ε, πίσω κατά, ε, κατά λίγο ως προς την ε, καινοτομία. Ο σύνδεσμός μας είναι ο υπεύθυνος από το Διαχειριστικό Συμβούλιο, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση. Merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και να ευχαριστήσω και τον οργανισμό για αυτή την εργασία αποτίμησης και ε, αντικτύπου. εξαιτία αυτού του απολογισμού και αποτίμησης μπορούμε να δούμε ποιος είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος τους πολίτες έτσι ώστε να έχουμε ένα, ε, μια επιστημονική υποστήριξη και πλατφόρμα ως προς την βιοπικιλότητα. Γι' αυτό ε, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ως προς την έκθεση του συναδέλφου Πάβαν Σούτπεκ μας αναφέρει ακριβώς ότι θα έχουμε απώλειες 50 ε, δις ευρώ μέχρι το 2050. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχουν γίνει αποτιμήσεις σε δύο θέματα. Καταρχήν, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες και οι οικονομικοί τομείς που είναι υπεύθυνοι για την απώλεια βιοπικιλότητας και έχουν γίνει αποτιμήσεις και ως προς τον έλεγχο των ε, κοινοτικών ενδιατημάτων που προστατεύονται έτσι θα μπορέσουμε να ορίσουμε τα καταλληλότερα μέτρα μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιοπικιλότητα και να προωθήσουμε και μια νέα, πολιτική, νέα αναπτυξιακή πολιτική για το 2020. Καλ Σλούτερ. and welcome. nice. Ναι, καλώς ήρθατε. Διάσα λίγο το πρόγραμμα εργασίας σας. Μου άρεσε το ότι αναφέρετε το ζήτημα της πράσινης οικονομίας και της αποτελεσματικής χρήσης πόρων. Γιατί μιλάτε και για συνεκτική πολιτική. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να πιστέψουμε πως η πράσινη τεχνολογία θα λύσει το πρόβλημα. Οπότε ποια κοινωνική πολιτική βλέπετε για το τι θα κάνουμε π.χ. με το χρόνο εργασίας, χρήση πόρων έτσι ώστε γιατί ε, π.χ. θεωρείται πως θα έχουμε με τα κέρδη αυτά περισσότερη καταναλωτική δύναμη ή περισσότερο χρόνο αναψυχής. Επίσης, τώρα είναι ο χρόνος της ε, βιοπικιλότητας ε, και θα είναι και το 2011 και ενδιαφέροντα και το φυλάδιο. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις ε, υπηρεσίες του οικοσύστηματος, ε, πώς θα λειτουργήσουν. Αν είναι να πιστέψουμε τον Ρόμπερτ Κωνσταντς από τη ΣΥΠΑ, που είναι ένας περιβαλλοντικός οικονομολόγος, το παγκόσμιο ΑΕΠ του περιβάλλοντος είναι δύο-τρεις φορές παραπάνω από τον ανθρώπινο ΑΕΠ. Οπότε θα καταδείξουμε φτωχότεροι αν το διαταράξουμε. Οπότε δεν είναι θέμα μόνο πόρων και αναψυχής, είναι και άλλες υπηρεσίες. Τι θα εξετάσετε λοιπόν, τι συμβουλές δίνετε στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εδώ συζητήθηκε μια αντίστοιχη έκθεση στην οποία είδαμε ότι εκφράζεται η λύπη που δεν έχει εκπληρωθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως συμφωνήθηκε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη στο Κέτερμπορκ το 2001. Δηλαδή να σταματήσει η απώλεια βιοπικιλότητας ως το 2010. Κατά τη γνώμη σας, κύριε κυρία Μαγκλέιντ, ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αποτυχία και τι στόχος πρέπει να μπει τώρα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ένα δεύτερο. επίση η έκθεση εκφράζει την ανησυχία για την έλλειψη προόδου σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον και ζητά από την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες. Τι δράσεις προτείνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για την προστασία του Ευρωπαϊκού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Και ένα τελευταίο, η ίδια έκθεση χαιρετίζει την αύξηση των δαπανών στο πρόγραμμα Life Plus κατά 8% σε σχέση με ε, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 αλλά υπογραμμίζει ότι αυτό το μέσο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό μόνο μέρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 0,2%. Ρωτώ λοιπόν τι προτείνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για την αύξηση του προϋπολογισμού του Life Plus και γενικότερα τι λέτε για την οικονομική υποστήριξη της προστασίας της βιοποικιλότητας. Thank you. Ευχαριστώ, Κρήτον Αρσένης. Thank you very much, Mr. President. Uh, I would like to welcome once more in, the, in this θα ήθελα να σας, να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά και επίσης θα ήθελα να ε, εκφράσω τη χαρά μου γιατί βλέπω ότι εστιάζουμε την προσοχή μας ε, σε ε, ένα, σε μια, μια νέα έκφανση των συζητήσεών μας εδώ. Ε, ο οργανισμός θέλει να επιδράσει στην βιοπικιλότητα, έτσι ώστε να έχουμε νέες πολιτικές ως προς την βιοπικιλότητα. Συνήθως έχουμε προβλήματα με τα στοιχεία και φαίνεται ότι έχουμε κατακαιρματισμένα στοιχεία και πολλές φορές αυτό αφορά και στοιχεία από τις μη κυβερνητικέ. Φαίνεται ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε τους δείκτες μας και ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μακλίτ πώς θα δημιουργηθεί μια επιστημονική εύρωστη βάση η οποία είναι ε, σημαντική για να φτάσουμε σε αυτές τις στοχοθετήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι έγινε το ΕΛΚ εξαϊλώθηκε, δεν υπάρχει πλέον αξιοσημείωτο. Οπότε εξακολουθούμε από αυτή την πτέρυγα να δίνουμε το λόγο. Γιούντιτ Μέρκης λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Μαγκλέιντ που ήρθατε και για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Σας έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, ένα θέμα που το συζητήσαμε ήδη, η εκπαίδευση, που είναι εξαιρετικά σημαντική. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας. Είναι το επόμενο θέμα βεβαίως. Τι θα γίνει με την ε, έλλειψη των πόρων, πώς θα μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα. Έχει την εντύπωση πως έχουμε σωστή πολιτική, είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα το κάνουμε αυτό ειδικά καθώς έχουμε και ένα... Αυτό είναι το σημείο 2 των προτεραιοτήτων της ε, Κομισιόν που είναι η αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα αναμένουμε μέχρι το τέλος του έτους την ανακοίνωση για τις πρώτες ύλες και του χρόνου από τον κύριο Ποτότσνικ την ανακοίνωση για το ίδιο θέμα. Και ο κύριος Γερμπάντη έκανε μία ερώτηση για την καινοτομία και ώρες, ώρες έχουν εντύπωση πως δεν βλέπουμε την ε, σχέση μεταξύ της ε, ε των ε, πόρων της σωστής χρήσης τους και του κλίματος. Π.χ. εγώ δεν βλέπω στις αξιολόγη, στην αξιολόγηση που λαμβάνουμε υπόψη το ότι οι πόροι σπανίζουν. Μιλάω π.χ. για το Desert Tech. Είναι ένα τεράστιο έργο. Έχουμε τους πόρους, έχουμε τα υλικά, να υλοποιηθεί ένα τόσο μεγάλο έργο. Εάν μιλήσουμε επίσης για όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα που απαιτούν τόσα υλικά, έχουμε υλικά για να κάνουμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Και τρίτον, ο αντίκτυπος της ε, οικονομικής κρίσης. Σήμερα συζητήσαμε για την καμπανία και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί πέρα, την κρίση με τα απόβλητα και έχουν εντύπωση πως λόγω της οικονομικής κρίσης κινδυνεύουμε να παραμελήσουμε πολλούς κανόνες περιβαλλοντικούς και την οδηγία για τα απόβλητα. Τις οδηγίες για τα απόβλητα, του χιτά και την εφαρμογή. Πώς θα διασφαλίσουμε λοιπόν το ότι παρά το ότι είμαστε σε ύφεση θα εξακολουθήσουμε να σεβόμαστε αυτές τις οδηγίες. Ευχαριστώ, Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Μακλέιτ, που ήρθατε εδώ. Την τελευταία φορά που ειδωθήκαμε ήταν στην Κοπενχάγη. Και αυτό που μπορώ να πω ήταν ε, ότι πάντα μας υποδεχτήκατε με μεγάλη θέρμη και ήσασταν ιδιαίτερα ε, αποτελεσματικοί σε όλα μας τα διαβήματα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω γιατί ήρθατε εδώ και μας δώσατε και ορισμένες πρόσφατες πληροφορίες. Αναφέρομαι στα, στις υπηρεσίες οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι τα συστήματα αυτά, πολλά από αυτά τα συστήματα έχουν αποδομηθεί. Άρα θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί γιατί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες από ορισμένα κράτη-μέλη ιδιαίτερα ε, από την ε, αντιπολίτευση σε σχέση με την γη, με τις ε, γέες, διότι το θέμα της υγιής αφορά και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και εδώ στην Ευρώπη. Άρα το θέμα της εξοικονόμησης των υδάτων είναι ύψης της σημασίας γιατί βλέπουμε ότι μειώνεται, μειώνεται ο υδροφόρος ορίζοντας, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Και αυτό που έχει σημασία είναι να εκμεταλλευτούμε πολύ σωστά αυτή την ε, δυνατότητα που έχουμε για να αποδώσει το σύστημα. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν είναι ύψης της σημασίας και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις γέες σαν ένα ε, οικολογικό σύστημα το οποίο δεν έχει μόνο τοπικό χαρακτήρα αλλά έχει και παγκόσμιους αντικτύπους, παγκόσμιο αντίκτυπο για την ε, διατήρηση και αποθήκευση του άνθρακα, για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και ούτω καθεξής. Πρόκειται για προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αποτιμηθούν από κοινού. Και θα πρέπει να κινηθούμε και εκτός Ευρώπης. Έχω πολλές αμφιβολίες για αυτή την παλινοδία ορισμένων κρατών μελών όσο αφορά ε, μία οδηγία που να αφορά τη, γη, τα εδάφη. Ελπίζω να σας απασχολήσει και αυτό το θέμα. Ναι, ε, το θέμα της οδηγίας για το έδαφος είναι ένα θέμα που ανακύπτει ε, κατά περιόδου. Η Λίντα Μέκατ. Λοιπόν, ο Βιτόριο Πρόντι μου θύμισε ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε ε, που μας ε, ε, φιλοξενήσατε στην Κοπενχάγη. Τότε καταλάβαμε κάπως ποια είναι η δουλειά σας. Το ερώτημα είναι αν γίνεται η σωστή χρήση της εργασίας του γραφείου σας και ε, ε, πρέπει, θα θέλαμε να ακούσουμε πώς εσείς αξιολογείτε τη χρήση της εργασίας σας από εμά, από την Επιτροπή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει διότι ε, θα πρέπει να, είσαστε, ε, να μην είστε ξεκάρφωτοι αλλά να συνεργαζόμαστε ως προς το τι προγράμματα αναλαμβάνετε διότι εδώ και έξι μήνες είχαμε συζητήσει ε, ότι θα βελτιωθούν οι σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να, είσαστε, να σας δοθεί μεγαλύτερη προβολή όχι μόνο από πλευράς περιβάλλοντος αλλά για πολλά θέματα νομοθετικά αυτή την εποχή ε, διότι ο οργανισμός σας ποτέ δεν είπε «Α, ασχολείστε ε, με αυτό». Δεν μας στείλατε κάποιο έγγραφο που να λέγει ότι ε, εκτιμάτε την εργασία μας. Επίσης, ε, θα ήθελα να ρωτήσω πώς χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δουλειά σας. Χρησιμοποιεί δικές σας πληροφορίες ή αναθέτει σε ανεξαρτήτους της μελέτης. Δηλαδή, μόνο το κοινοβούλιο κοφεύει. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα διότι οι περισσότεροι βουλευτές τους οποίους ακούω είναι η τρίτη μου θητεία στην Ευρωβουλή αλλά ε, ε, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που θα έπρεπε να απευθυνθώ εάν θέλω κάτι από τον οργανισμό σας διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι προβαίνουν σε έρευνα και καλό θα ήταν να ε, κατανοήσουμε όταν υπάρχει ένα συγητής για ένα μείζον θέμα. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δίνετε ε, και τι πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικά αυτά. Πολύ σωστές ερωτήσεις και ο τελευταίος ο, μιλητής είναι ο Πας Έικουτ. Θα είμαι σύντομος. Πάντοτε είναι χαρά που έρχεστε εδώ και νομίζω ότι αυτό έχει σχέση με ό,τι είπε η Κιλίντα Μακάβεν. Αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας διότι ε, ξέρετε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, ξέρετε Ξέρουμε ότι η ΕΕ προσπαθεί να παρακολουθήσει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσεγγίζει τους στόχους που έχει θέσει και ιδίως για τους στόχους του 2020. Αλλά στην έκθεση αυτή αναλύεται επίσης και τις δυνατότητες αυξήσεως των φιλοδοξιών σε επίπεδο κρατών μελών, πέραν δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Επιτροπή λέει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το 30% Οπότε τι σημαίνει αυτό για τα κράτη-μέλη. Μήπως ε, ε, το φθινόπωρο θα μπορούσαμε να έχουμε μία έκθεση που να αναφέρεται εις ε, το θέμα των κρατών μελών διότι μέχρι στιγμής έχει υπάρξει διξα... δισταγμός να αναλυφθούν όλα αυτά. Ε, νόμιζα ότι σας είχα ξαναδεί. Έχετε πολλές ερωτήσεις αλλά δεν θυμήθηκα ότι σας είχα δει το Δεκέμβριο στην Κοπενχάγη. Σας ευχαριστώ λοιπόν και σας δίνω το λόγο. Καλά θυμάστε κύριε Πρόεδρε. Είχα ξαναέρθει. Τέλος πάντων να ασχοληθώ τώρα με τις ερωτήσεις. Όσον αφορά την μίεση και την πιθανή αύξηση μετά ξανά. Έχω την έκθεση που βγάλαμε σήμερα και έχει και ανακοίνωση που μας δίνει μια καλή ιδέα του που από πού προήλθαν αυτές οι μειώσεις θα δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον, έχουμε μια μετάβαση στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στις πηγές ε, καυσίμων δηλαδή που πάνε προς τα εκεί και αυτή είναι η συστημική αλλαγή. Αλλά υπάρχουν πράγματι στοιχεία ότι σε κάποιες χώρες, π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ιταλία ε, υπάρχει μετάβαση σε βιοκαύσιμα. Οπότε ήδη υπάρχουν νέες ροές που δεν νομίζουμε πως θα εξαφανιστούν. Οπότε υπάρχουν καλά σημάδια από τον τομέα της ενέργειας. Μπορείτε να πείτε πως το γεγονός ότι στη Γερμανία η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε από θερμική ενέργεια και ε, αυξήθηκε η πυρηνική, μπορεί να μην είναι αυτό που θέλατε, αλλά αυτό συνέβη. Υπήρχε μια ενδιαφέρουσα μείωση από την παραγωγή νητρικού οξέως, ειδικά από την παραγωγή στα Ολλανδικά εργοστάσια. Οπότε βλέπουμε σημεία τα οποία δεν περιμένουμε να ξανανεύουν οι εκπομπές. Και κάποια άλλα, π.χ. παραγωγή σιδήρου, χάλιβα και μεταφορές. Από την άλλη βεβαίως υπάρχουν και αυξήσεις που ε, αντικαθιστούν λίγο αυτές τις μειώσεις, π.χ. υπηρεσίες νοικοκυριά αυξάνονται, πρέπει να προσέχουμε εκεί. Επίσης όταν κυμαίνονται οι τιμές ε, προσαρμόζονται ανάλογα και τα αποθέματα καυσίμων στις χώρες, οπότε αυτό μας μπερδεύει, πρέπει να προσέχουμε γιατί καμιά φορά υπάρχουν μεγάλες διακοιμάσεις, αλλά έχουμε και με κάποιες μειώσεις στον κλωριοθωράνθρακα ε, και αντικαταστήτη από άλλα αέρια στα ψυγεία και τα κλιματιστικά, οπότε πρέπει να προσέχουμε και εκεί πέρα. Σα παρακαλώ λοιπόν να διαβάσετε την έκθεση, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αρχίζει να κοιτάει τις μελλοντικέ τάσει. Τώρα να έρθουμε στην καινοτομία. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι πως σε άλλε χώρε ε, στη ΣΥΠΑ και σε έναν βαθμό ε, και στην Ιαπωνία, ε, έχουμε έντονη καινοτομία επίπεδα επένδυση ρεκόρ που δεν υπάρχουν εδώ πέρα στην Ευρώπη, οπότε θέσει το δάκλειο από τον τύπο των Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ε, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της ύφεση να μην ε, μειωθεί η επένδυση στην καινοτομία, ειδικά στο πρασίνισμα, όπως λέμε, της οικονομίας. Τώρα, όσον αφορά την βιοπικιλότητα, ποιοι είναι οι τομείς υπεύθυνοι. Εγώ θα έλεγα γεωργία, χωροταξία που κυριολεκτικά εξαπλώνονται οι πόλεις και μεταφορές. Αυτά είναι τα τρία βασικά στην ξηρά και βεβαίως στη θάλασσα αλληλεία. Αλλά θα συνεχίσει αυτή η τάση στα περισσότερα αλλιεύματα. Τώρα, πώς ξεφεύγουμε από αυτό, ρωτήσατε. Συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν και εσείς αναφέρατε τη βιοπικιλότητα. Κοιτάξτε, χρόνο με το χρόνο η σχέση μας με την Κομισιόν βελτιώνεται και οπωσδήποτε ε, στο διάλογο με την Κομισιόν νομίζω πως έχουμε πολύ καλή σχέση εργασίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πολλές από τις εκθέσεις και τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουμε αποτελούν τώρα στοιχεία για το πώς θα έχουμε πραγματικά αυτή την πλατφόρμα ε, αποτελεσματική χρήσης ενέργειας και πώς θα συνδεθεί με την βιοπικιλότητα. Οπότε αυτό το σύστημα εδώ πέρα ήταν μια προσπάθεια δική μας και της Κομισιόν και του Κοινού Κέντρου Έρευνα. Οπότε ήταν μια συνδυασμένη προσπάθεια όλων μας τις τελευταίες 12 εβδομάδες για να δώσουμε μια μεγάλη όθηση στο να μαζέψουμε πληροφορίες και έτσι επανερχόμαστε στους τομείς. Ε, όταν ε, θέσαμε στόχους, αυτή τη φορά είχαμε την ιδέα μαζί με την Κομισιόν να θέσουμε υποστόχους προς τους τομείς εκείνους που εμείς θεωρούμε πως επιδρούν στη βιοπικιλότητα. Και αυτή είναι στόχοι που δεν είναι εκτός τη βασικού, της βασικής δουλειάς αυτών των κλαδίων. Δηλαδή π.χ. σαφώς αλληλεία, αλλά να δούμε και τους θαλάσσιους τροφικούς δείκτες, όχι μόνο αναείδος, αλλά να το δούμε από τα μεγάλα αρπακτικά προς τα κάτω και αυτό είναι το σκεπτικό της αποκατάστασης και επανερχόμαστε σε αυτό γιατί αναγνωρίζουμε και αυτό είναι κάτι που ξέρουμε τώρα πως ο ευτροφισμός στο θαλάσσιο περιβάλλον επιτείνεται όταν δεν υπάρχουν όλα τα επίπεδα. αυτό γίνεται για τη Βαλτική, γιατί έχουμε ακριβώς αυτή την άνθηση των φυκιών, γιατί έχουμε χάσει πολλές, πολλά από τα κομμάτια της αλυσίας, πολλά από τα μεγάλα αρπακτικά. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε στο παρελθόν, στην στο γλυκό νερό μάλλον, με συγχωρείτε, ε, στην ξηρά μεταφέρεται τώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε επανερχόμαστε σε τομιακούς ε, στόχους, οπότε μιλάμε συνολικότερα για οικοσυστήματα και όχι μόνο για τα εμπορικά είδη. Το ίδιο και με τη γεωργία. Βλέπουμε συγκεκριμένα ωφέλη όταν ε, κοιτάμε τη γεωργία πλευράς χρήσης γης και αλλαγής χρήσης γης, να περάσουμε από την εκτατική ε, καλλιέργεια αρωτρέων γεών σε μια πιο επικεντρωμένη καλλιέργεια, να δούμε επίσης πώς γίνεται η χρήση του νερού και να έχουμε κεντρικούς στόχους για να δούμε ένα ποσοστό μετάφερες νερού για να έχουμε μια ενισχυμένη εικόνα. Οπότε έχουμε αυτούς τους υποστόχους που αναπτύσσονται μαζί με τους συναδέλφους στην Κομισιόν και αυτό επανέρχεται στην καθημερινή μας δουλειά με τα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε υποστόχους στη δασοκομεία, γεωργία, αλληλεία κτλ. Βεβαίως, πολεοδομία, μεταφορές και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε κάποια ιδέα λόγω της κατακαιρματισμού από την εξάπλωση των πόλεων. Επίσης είπατε πως υπάρχουν κενά πράγματι στις περιοχές οποίες διαχειριζόμαστε και βλέπουμε πως αν ε, θέλετε οι εισβολές στις περιοχές Natura 2000 είναι ένα από τα προειδοποιητικά καμπανιάκια. Οπότε εκεί πέρα το πρόγραμμα GMS θα μας βοηθήσει γιατί έχουμε πάρα πολύ γρήγορη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε πλέον πέντε χρόνια. Ελπίζουμε να έχουμε ενημέρωση κάθε χρόνο. Οπότε θα μπορούμε να έχουμε πολύ πιο γρήγορα ε, μηνύματα όλοι μας για το που βλέπουμε κινδύνους στις άκρες των προστατευμένων περιοχών, κυρίως στην ξηρά. Οπότε η δυνατότητα ενημέρωσης ε, για την γνώση που θα έχετε και η κατανόηση βεβαίως θα είναι πολύ καλύτερη οπότε αναμένουμε βεβαίω και καλύτερη επιβολή και σε αυτό θα πιέσουμε. Κάρλ για την ιδέα σας για την αποτελεσματική χρήση πόρων αυτό είναι πράγματι σωστό, είναι καλό ε, να μου λέτε ότι αυτό θέλετε αλλά για να επανέλθω στο πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή και πώς θα συνδεθούν οι υπηρεσίες ε, οικοσυστημάτων. Κάνουμε πολλή δουλειά στην οικονομική πτυχή, την αξιολόγηση. Σήμερα μάλιστα βγάλαμε και άλλη μια έκθεση για να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα που λέγεται τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοπικιλότητας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη γιατί λέει πως είναι ε, πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις, πρέπει να δούμε το τοπικό πλαίσιο και άρα επανερχόμαστε στο πώς αντιμετωπίζουμε τις υπηρεσίες κοστιμάτων. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα είναι μία πρώτη προσπάθεια, το βλέπετε στον πίνακα αυτό, στο πίσω μέρος, όπου εξετάζουμε τις υπηρεσίες κοστιμάτων που έχουν βλεπτεί σε διάφορα ενδιαιτήματα ανά χώρα. Οπότε βλέπετε πως προσπαθούμε πραγματικά να διαρθρώσουμε και να δούμε ποιες οι υπηρεσίες από αυτές χρειάζονται την προσοχή μας και μετά θα αναπτύξουμε δείκτες. Αλλά όπως σας είπα προσπαθούμε να διευρύνουμε την συζήτηση για να συμπεριλάβει μια ανάλυση κύκλου ζωής που θα πηγαίνει πέρα από τη βασική χρήση πόρων όπως γη και νερό και να δούμε τις υπηρεσίες κοστιμάτων που χρειάζονται για να δημιουργήσουμε μια οικονομία αποτελεσματικής χρήσης πόρων. Μετά βλέπουμε ε, φόρους βεβαίως, ε, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το πώς θα είναι η κατανάλωση, κίνητρα και αντικίνητρα και βλέπουμε εκεί πέρα καλές ιδέες από άλλα μέρη του κόσμου που δεν είναι μόνο η, η τιμή αυτή η οποία αλλάζει την κατανάλωση. Το νερό είναι ένας πάρα πολύ καλός δείκτης ότι βεβαίως η τιμή δεν είναι πάντα η απάντηση. Π.χ. στην Αυστραλία και στη ΣΥΠΑ σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες είναι η αηφορία της προμήθειας νερού που άλλαξε τη συμπεριφορά και όχι απόλυτη τιμή. Οπότε πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτοί στην Ευρώπη και να δούμε άλλες βέλτιστες πρακτικές από άλλα μέρη του κόσμου όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά κάποιες καλές ιδέες και ε, ευχαριστώ μπορούμε να έχουμε αυτές τις ιδέες και στην Ευρώπη για να δούμε πώς θα έχουμε αυτές τις υπηρεσίες εδώ πέρα. Τώρα για την θάλασσα. Είχαμε μια καλή συζήτηση στην Πράσινη Εβδομάδα για το πώς μπορούμε να δούμε το ευρύτερο ζήτημα. Έχουμε δύο μόνο θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές από 1500 θα μπορούσαμε δυνητικά να έχουμε. Οι περισσότερες βεβαίω είναι κοντά στην ε, ακτή, αλλά πρέπει να δούμε και της, ε, υπερ τις υπερπόντιες κτήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς 10% των κοραλιογενών υφάλων βρίσκονται σε ευρωπαϊκή επικράτεια, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε θεωρώ πως ε, πρέπει να δούμε πώς θα επιτηρήσουμε, θα παρακολουθήσουμε αυτές τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, γιατί αν σκεφτούμε τις αποτυχίες, είναι ε, το ότι δεν ξέρουμε αρκετά για την αλληλεπίδραση μεταξύ τομέα και συγκεκριμένου ενδιατήματος. Τώρα για το Life και το IF Plus δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα ήθελα προφανώς περισσότερες επενδύσεις, αλλά πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά την ισορροπία μεταξύ πρασινίσματος οικονομίας ε, και ζητημάτων που είναι καθαρά περιβαλλοντικά. Τώρα για τους δείκτες, νομίζω πως έχουμε για τους δείκτες βιοπικιλότητας η κατάσταση βελτιώθηκε ακόμα και σε σχέση με πέρσι και νομίζω πως το ταρακούνημα που είχαμε όταν ο τότε επίτροπος ο κύριος Δήμας προείδε ότι δεν θα επιτύχουμε τον στόχο, νομίζω μας ανάγκασε να πούμε πως δεν έχουμε αρκετούς δείκτες για να δούμε όλο αυτό το φάσμα ζητημάτων. Οπότε τις τελευταίες αυτές 12 εβδομάδες πραγματικά επιταχύναμε και η επιστημονική κοινότητα νομίζω και εμείς ε, καταφέραμε να βρούμε κάποιους καλύτερους βασικούς δείκτες οι οποίοι βεβαίως είναι εύρωστοι, μπορούν να βελτιωθούν πάντα αλλά μας δίνουν μια βάση για την εκπαίδευση. Συμφωνώ πλήρως. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο που θα διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές αυτές ε, διαδικασίες στα κράτη-μέλη και το λέω αυτό γιατί θεωρώ πως υπάρχει μια ιστορία που πρέπει να πούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο που δεν περνάει στα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Θεωρώ πως ειδικά η δική μου υπηρεσία πρέπει να φτιάξει τέτοιες περισσότερες ιστορίες, αν θέλετε, τα επιχειρήματα, το ευρωπαϊκό αποτύπωμα ή το υδάτινο αποτύπωμα ή ό,τι άλλο. Να γίνει δηλαδή σαφές ότι σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να μάθουμε κάτι και μετά να κλιμακωθεί και να αποκλιμακωθεί στο παγκόσμιο και το εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε όταν μιλάμε για πραγματική ε, σπάνιδα να δούμε πώς ε, βασιζόμαστε στους παρθένους πόρους εντός των συνόρων της Ένωσης. Νομίζω πως ε, μια καλή αρχή είναι η δουλειά και της δικής μας υπηρεσίας και με το Διεθνές πάνελ για τη χρήση των πόρων, των μετάλλων, ειδικά για τις σπάνιες γέες και αυτά που βρίσκονται στο περιοδικό πίνακα μαζί με το σιδηρομετάλλευμα, όλα αυτά που εξαρτώνται δηλαδή από μεταλλεία στην Αφρική, αλλά και εξαρτώνται και οι δικές μας βιομηχανίες από αυτά γιατί δεν ανακυκλώνουμε αρκετά. Οπότε θα πρέπει να έχουμε καλύτερη ανακύκλωση και μετά θα ήταν τελείως διαφορετική η συζήτηση για τα μέταλλα, τα μεταλλεύματα και όλα αυτά. Τώρα, πρωτοβουλίες σημαίες, αν θέλετε. Ναι, να δούμε ε, τις ε, πρώτες ύλες, ε, καλύτερη χρήση μέσω της κοινοδομίας και βελτίωση αυτών που έχουμε. Π.χ. συσκευασία μπορούμε να την ξαναδούμε. Είναι μεικτή η εικόνα. Αν κάναμε καλή δουλειά στην ανακύκλωση των συσκευασιών θα βελτιώναμε την αποτελεσματικότητα των πόρων. Για τον Desert Tech δεν θα περάσω στις λεπτομέρειες, μπορούμε να το δούμε με διάφορους ε, τρόπους, ε, χωρίς αυτό να σημαίνει πώς θα κινητοποιηθούν γρήγορα μεγάλες ποσότητες υλικών, αλλά πρέπει να είναι σαφές πως κάθε αξιολόγηση αντικτύπου από εδώ και μπρος θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει το πού βρίσκονται τα υλικά, πού είναι η καινοτομία, από πού θα είναι η κινητοποίηση για να γίνουν όλες αυτές οι πολιτικές και πολύ περισσότερο βεβαίως από όλα τα άλλα το νερό και η σπάνης αυτή των πόρων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε στο πρόγραμμα εργασίας. Νομίζω λοιπόν πως ε, όταν κάνουμε αυτές τις ε, εξελογές που μπορούμε να ταιριάξουμε και αυτά τα πράγματα εκεί μέσα. Επίσης εφαρμογή όπως ε, συζητήσαμε και νωρίτερα είναι πάντα ένα θέμα οπότε το να δίνουμε προτεραιότητα σε κάποιους τομείς είναι χρήσιμο για το λόγο και μόνο ότι βεβαίως θα ενσωματωθεί και στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και σε άλλους ε, τομείς της πολιτικής και έτσι θα έχουμε μια συνακτική ε, πολιτική και βλέπω πως με το πάνελ αυτό το οποίο θέλει να δημιουργήσει η Κομισιόν για την αποτελεσματική χρήση των πόρων και το 2020 θα έχουμε μια συνεκτική πολιτική. Για τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, Βιτόριο, βεβαίως θα α, έλεγα πως πρέπει πάντα να λέμε πως εάν εστιάσουμε πάρα πολύ σε ένα σημείο κάτι άλλο θα μας ξεφύγει και αυτό βέβαια για το έδαφος. Εγώ είμαι υπέρ του να παραμείνει η οδηγία εδαφών στο σωστό το δρόμο γιατί βεβαίως εάν χάσουν τα εδάφη τη δυνατότητα να παγιδεύουν διοξείδιο του άνθρακα ε, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Τέλος για να επανέλθουμε και στην αρχή, το μείον 30% είναι ένας πολιτικοποιημένος τομέας όπως ξέρετε. Ε, κούτσα κούτσα εκεί πέρα με τους συναδέλφους στην Κομισιόν προσπαθούμε να μην ε, γίνουμε πάρα πολύ πολιτικοποιημένοι. Μπορούμε να ακολουθήσουμε πολλούς δρόμους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε ακόμη πιο επιθετικούς στόχους. Αλλά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταματήσει η τεχνική συζήτηση και να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις. Γιατί καμιά φορά, αν δούμε το τι γίνεται ανά τον κόσμο όσον αφορά την καινοτομία, νέα υλικά, ενέργεια κτλ. Αυτό το οποίο με ρωτάνε είναι αν κάποιος θέσει τον πύχη θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί δεν υπάρχει μία τεχνολογία που θα φέρει την αλλαγή. Είναι ένα συστημικό ζήτημα αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε να εξετάζουμε νέες τεχνολογίες από παραπάνω από μία πτυχές. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα ζήτημα εκπομπών, είναι να κάνουμε μία ανάλυση κύκλου ζωής στα πάντα. Στην επίδραση για τους σπόρους, για τη γη, για το νερό, οπότε πρέπει, ε, η πρωτοποίησή μου είναι, εντάξει να μην λέμε 50-80% μείωση, δεν θα είναι μόνο από την πτυχή των ε, αερίων ε, του θερμοκηπίου, γενικά η επίδραση στο περιβάλλον. Αυτό κάνουμε εμείς στην έκθεσή μας σε σχέση με τις μεγάλες τάσεις στον κόσμο. Οπότε κάποιες από τις απαντήσεις οπωσδήποτε υπάρχουν και θα τις λάβετε σε, σε τέσσερις μήνες περίπου. Δεν ξέρω, μπορεί και ίσως νωρίτερα. Ευχαριστώ κυρία Μακλέιν για αυτή τη συζήτηση. Είναι προφανές ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος και τα μέλη της αποδίδουν μεγάλη σημασία στο να έχουμε μια στενή επαφή. Βλέπουμε πόσο σκληρά εργάζεστε στην Κοπενχάγη, πόσα πολλά στοιχεία προσπαθείτε να συγκεντρώσετε για να έχει κανείς μια σωστή εικόνα και τον προβλημάτων προβλημάτων και της στρατηγικής για τη σωστή επίλυση των ε, προβλημάτων. Αναφερθήκαμε σε τρία-τέσσερα σύνολα προβλημάτων που μας ενδιαφέρουν πολύ, την κλιματική προστασία, την βιοπικιλότητα, άλλο μεγάλο θέμα και την αποδοτικότητα των πόρων. Όσον αφορά την την ε, οδηγία για τα απόβλητα των ηλεκτρικών συσκευών είναι κάτι που μας απασχολεί και υπάρχουν και άλλα θέματα όπου ζητούμε να καταρτιστεί ένα πλαίσιο κανόνων ε, και αυτή η Επιτροπή είναι πολύ ενεργή στην επιζήτηση αυτών των στόχων κατά τρόπον ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων. Προσβλέπω στην ανακοίνωση της Επιτροπής που θα δημοσιευθεί σχετικά με αυτό το θέμα και όπου θα αποτελέσει τη βάση της περαιτέρω εργασίας μας. Σας ευχαριστούμε, ελπίζουμε να σας ξαναδούμε ε, σύντομα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέχασα, είναι ένα πρακτικό θέμα, υπάρχουν πάντε συνάδελφοι ε, εδώ οι οποίοι ίσως κάθονται στο βάθος. Γιωχάνες μπορείτε να σηκώσετε το χέρι σας. Ο Γιωχάνες είναι πάντοτε εδώ, είναι από την Επιτροπή μας, μπορείτε να τον προσεγγίσετε διότι προσπαθούμε να παρακολουθούμε τι χρειάζεστε και ειλικρινά πιστεύουμε ότι εάν δεν προχωρά σωστά η συνεργασία μας μαζί σας, πέστε μάστε το και θα κοιτάξουμε να τη διορθώσουμε. Και το λέω αυτό διότι μιλώ με πολλούς συναδέλφους συχνά στο τηλέφωνο και γι' αυτό θα ήθελα να μπορώ να στείλω και την ίδια ε, πρόσκληση προς άλλους. Ευχαριστούμε. Καλό είναι να ξέρουμε ποιοι είναι οι συναδελφοί σας κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να τους προσεγγίζουμε όποτε χρειάζεται. Λοιπόν, αύριο 9 το πρωί συντονιστές και 10 η ώρα συνέχεια της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και έληξε η συνεδρίαση.